και μπορείτε να το δείτε ή στο κομπιούτερ σας ή στην τηλεόραση. Τέλος πάντων θα σας ενημερώσουμε πού θα γίνει η προβολή. Ε, η Ιζαμπελ Ντιρόν και εγώ ήμασταν στη Βενετία και είδαμε αυτές τις τρεις ε, ταινίες ε, μαζί με τους... που ήταν εκεί. Επίσης ε, συζητήσαμε με πολλούς νέους ενδιαφερόμενους για τον κινηματογράφο. Τους είχαν προσκαλέσει στο φεστιβάλ της Βενετίας. Συζητήσαμε το μέλλον του κινηματογράφου και 27 ε, χώρες είχαν εκπροσωπηθεί στην Βενετία και διαπιστώσαμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ καλό και λειτουργικό ευρωπαϊκό δίκτυο κινηματογράφου και αυτές οι ταινίες έχουν γυριστεί από νέους ανθρώπους και αυτοί θα μείνουν σε επαφή μαζί μας ε, και επειδή υποστηρίζουμε ιδιαίτερα τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο πιστεύω ότι εδώ έχουμε επιτύχει να ε, τους εμπνεύσουμε με την ευρωπαϊκή ιδέα του, του υψηλού επίπεδου κινηματογράφου. Ε, ήταν λοιπόν πάρα πολύ ωραία και ζουμερή αυτή η επίσκεψη. Επίσης, ε, του χρόνου στη Γερμανία, εκτός από τις 27 χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καλέσουμε και νέους ε, παραγωγούς και σκηνοθέτες από τις Βαλκανικές χώρες. Θα έχουμε 34-35 νέους κινηματογραφιστές που θα συναντηθούν λοιπόν του χρόνου. 27 συν άλλες χώρες, άλλες 5-6 χώρες στις 15-16 ε, Νοεμβρίου, πριν την απονομή του βραβείου Λουξ, θα κάνουμε μία συνάντηση με δημοσιογράφους από όλες τις χώρες και ένα σεμινάριο θα διοργανώσουμε μαζί με τους παραγωγούς, τους κοινοθέτε των ταινιών αυτών, όλους δηλαδή που έχουν συμπράξει στη δημιουργία αυτών των ταινιών. Θα συζητήσουμε τον κινηματογράφο, τις ταινίες και Α, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση του Μπόρι στην ε, Ολομέλεια. Αύριο θα λάβετε όλες τις πληροφορίες στην πρόσκληση. Σας παρακαλώ να διαδώσετε το μήνυμα στους συναδέλφους για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ε, διαδικασία επιλογής του βραβείου. Η κυρία Μπενερά Πατού έχει μία ερώτηση και μετά θα αρχίσουμε ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση σε σχέση με την επιλογή των νέων στη Μόστρα. Πώς θα γίνει η επιλογή. Οι νέοι που θα έρθουν προσκαλούνται από το ΣΥΝΕ Europe, ε, Ευρώπη. Αυτοί τους επιλέγουν, ε, δημοσιεύουν μια προκήρυξη, εξετάσουν τις αιτήσει και επιλέγουν ποιους θα προσκαλέσουν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τι έχει κάνει, το βιογραφικό του, τι, τι λοιπά. Ε, εμείς ε, δεν έχουμε καμία επιρροή στην επιλογή, ε, το ΣΥΝΕ Europe, Cine Europa. Τους διαλέγει. Η ημερήσια διάταξη τώρα και αρχίζουμε με την ψηφοφορία για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πάρα πολύ απλό. Σας παρακαλώ ψηφίστε υπέρ, υπέρ του σήματος. Ωραία. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Α, δύο παραπάνω είναι από το ΕΛΚ. Είναι δύο πλεονάζοντες. Είναι εντάξει τώρα. Ωραία, ωραία. Καλή οργάνωση. Μπράβο. Λοιπόν, Ωραία, είσαστε παρόντες, δεν θα ψηφίσετε, ε, δεν μπορείτε να ψηφίσετε, αλλά σας συγχαίρω που είσαστε παρόντες. Λοιπόν, υπέρ, ψηφίζουμε υπέρ του σήματος, παρακαλώ. Κατά, αποχές, κανείς. Πολύ ωραία. Ομόφωνα εγκρίσκει, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κυρία Παγιαδέλη και τους κοιόδης συζητητές. Προχωρούμε στην έκθεση. Ναι, δεν ήταν τόσο εύκολη. Έγινε μεγάλο έργο που σκληρή δουλειά έγινε και εντάξει, τα καταφέραμε. Ε, το Ευρωπαϊκό Σχηματογράφο στην ψηφιακή εποχή. Έξεση του κυρίου Μπόρις. Α, περιμένει το μωρό του, το μωρό του. με τη γυναίκα του. <laughs> Περιμένει τον τοκετό. Δεν μπορεί να είναι εδώ παρόν. Έχουμε κατανόηση και έχουμε τον κατάλογο ψηφοφοριών. Το 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές Α, άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται 15 προς 8. 39. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. 38 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 40 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 41 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36, 46 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ κατά. Α, καταπίπτει. Ναι. 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ, ε, συγγνώμη, 63 κατά αποχές δεκτή, 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 69 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονική παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία έληξε η ψηφοφορία δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 16 προς 12. 73 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 76 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 77 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 78 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 79 υπέρ, κατά, αποχές, α, ηλεκτρονική παρακαλώ. Άρχεται, πέρας. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Απο, αποχές. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή.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 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά 95 κατά αποχές δεκτή. 96 ε, καταπίπτει. 97 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 97 παρακαλώ. Άρχεται, πέρας, Δεκτή. 98. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 99. Καταπίπτει. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 δεκτή 109 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 111 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 114 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 115 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 118 Α, η, η, η έκδοση αναφοράς είναι η γαλλική, στη γαλλική γλώσσα. Υπέρ, κατά. Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 120 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 14 προς 13, δεκτή. 121 υπέρ κατά αποχές έλεγχος πάλι. Άρχεται ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 122. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 123. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 124. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 125. Τίποτα. Δεν επηρεάζει το είναι αγγλική έκδοση. Λοιπόν, 127 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 128 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 129 διαχωρισμό στην ψηφοφορία πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές Έλεγχος του δεύτερου μέρους παρακαλώ της 129. Άρχεται η ψηφοφορία, έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές. Δεκτή, 132 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 133 διαχωρισμός της ψηφοφορίας. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτω. 135 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία, έληξε ψηφοφορία. 16 προς 11 απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 134, α, 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 138 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 139 υπέρ κατά, απο, κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 141 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέραση ψηφοφορίας 15 προς 14 δεκτή πάμε στο 149 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Απο, απορρίπτεται. 151, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 152, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 153 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 159 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 160 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 161 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 162 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 163 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 166 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 168 υπέρ κατά αποχές έλαφος. Έλαφος παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία, έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 170 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 171 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 172 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 173 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 175 δεκτή, 176 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 177 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 179 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 180 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 181 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 182 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 183 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος παρακαλώ την 183. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 185 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 189 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 190 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 191 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 192 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εγώ λέει χαλάω τη φωνή μου, λέει η πρόεδρος. <laughs> 95 δεκτή 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές α καταπίπτει η 6 ναι ναι εντάξει 7 7 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ Δεκτή. Εννέα υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Δέκα υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Έντεκα υπέρ Δεκτή. δώδεκα, Υπέρ κατά αποχές δεκτή. δεκατρία, Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. δεκατέσσερα, Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 19 υπέρ, κατά, έλεγχος παρακαλώ, τη 19. Απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 27 υπέρ κατά δεκτή, 28 υπέρ κατά δεκτή, 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στη γνωμοδότηση ΙΜΚΟ. Μπορούμε να τις πάρουμε όλες μαζί σε γκρουπ, 1, 2, 3, 4. Όχι. Θεέ μου λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, πά. Ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή, δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή, τρία δεκτή, τέσσερα υπέρ κατά δεκτή. Ε, ναι. Τώρα, Λοιπόν, 5 υπέρ κατά δεκτή, 6 υπέρ κατά είχε δεκτή, 7 ναι, δεκτή, 8 ε, δεκτή και λοιπά και λοιπά, 9, 10 δεκτή, 11 δεκτή, 12 δεκτή, 13 δεκτή. Μάλιστα, θέ μου. <laughs> Και τώρα η τελευταία ψηφοφορία παρακαλώ για ολόκληρη την γνωμοδότηση υπέρ, κατά. 28 προς 0. Μπράβο, μπράβο, είναι απίστευτο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχα... ευχαριστούμε τον κύριο Μπόρις, ελπίζω να είναι καλά και το μωρό. Ωραία, προχωρούμε στην κυρία Χάνιμπολ. the floor on compromise one and 45. Why not? Any So, uh, I was told I should give the floor to... Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Χάνιμπολ και τον κύριο Σκουρία για τον συμβιβαστική ένα. Ε, ε, τι γίνεται. Κοιτάξτε, λέει η κυρία Χάνιμπολ. Πόσο γνωρίζω, θα πρέπει να αρκεστούμε στον κατάλογο ψηφοφορίων. Ξέρω ότι ο κύριος Σκούρια έχει μία τροπολογία που θεωρεί ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στον συμβασμό. Πρόκειται για τον Σύμβασμο υπαριθμών 1 και εάν περάσει, θα περάσει με την κανονική διαδικασία. Εάν δεν εγκριθεί, τότε θα ψηφίσουμε επί των μεμονωμένων τροπολογιών. Δηλαδή θα αρκεστούμε στην κανονική διαδικασία. Σκούρια με την τροπολογία 45 που υπέβαλα. Υπέβαλα μία προσθήκη σε σχέση με το κείμενο που προέβλεπε ε, τις ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, δηλαδή να μιλάμε για μία κοινωνία η οποία θα βασίζεται στην ισότητα, στη μη διάκριση αλλά και στην αξιοκρατία. Γιατί και η αξιοκρατία είναι σημαντική σε μια κοινωνία. Γι' αυτό ήθελα να συμπεριλευθεί. Οι σοσιαλιστές μου είπαν ότι είναι δύσκολο κάτι τέτοιο. Ελπίζω όμως παρόλα αυτά να μπορέσει να συμπεριληφθεί. Μάλιστα. Δεν θα αρχίσουμε συζήτηση. όσοι θέλουν να ψηφίσουν τη 44 πρέπει να καταψηφίσουν τη συμβιβαστική 1. Αλλά ο κύριος Σκούρια είναι επιφυλακτικός. Τι θέλετε να κάνουμε. Εσείς δώστε το σήμα με το χέρι σας, είναι δική σας η τροπολογία και εσείς θα αποφασίσετε εάν θα υπερψηφίσετε ή καταψηφίσετε τη συμβιβαστική. Το αφήνω σε εσάς. Λοιπόν, αρχίζουμε. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές... Α, έλεγχος παρακαλώ. Zu 11, angenommen. Δεκτή, δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Αρχίζει, άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 από την απασχόληση. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτό. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 33 υπέρ κατά αποχές ξανά. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2 της απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 35 υπέρ. Α, καταπίπτει, καταπίπτει. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, πρέπει να ελέγξουμε. Έληξε ψηφοφορία. 17 Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 40 παρακαλώ. Ε, έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. 20 προς 8 δεκτή. Οπότε προχωράμε στην 48 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 49 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 52 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε παρακαλώ. 52. Έληξη ψηφοφορία. 14 προς 15 απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 55 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 56 υπέρ, κατά, αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Πάμε στην 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ναι. Ωραία. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> Δεκτή. 68. Υπέρ. Α, ε, συγγνώμη, συγγνώμη, 74. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 75. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 76. Υπέρ κατά αποχές. Α, να ελέγξουμε την 76. Ξανά. Δεν Κάποιος δεν μπορούσε να ψηφίσει. Δεκτή πάντως. Η 76. Πάμε στην 79. υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 89 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, 89 παρακαλώ, ε, τη ψηφοφορίες. Δεκτή, 90 υπέρ Α, καταπίπτει. 91 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 92 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 94 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές δεκτεί. 98 υπέρ κατά αποχές δεκτεί. 99 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Έλεγχος παρακαλώ στην 99. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτεί. 100. Δεκτεί, δεκτεί. 102. 102. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α, έλεγχος παρακαλώ. Έλεγχος στην 106. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τοπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 119 υπέρ κατά ένα λεπτό, 119 υπέρ κατά Αποχές δεκτή. Προφορική τοπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Οι σοσιαλιστές ψηφίζουν μαζί μας. Πού πάμε τώρα. Στην 11. 11. Εμπλουά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε το δεύτερο μέρος, το δεύτερο τμήμα παρακαλώ, της 126. Έγινε δεκτό, ε, δεκτό, 18 προς 10, 120, 127, 128, υπέρ, κατά, δεκτό. 129 υπέρ κατά δεκτό 130 υπέρ κατά αποχές δεκτό 131 υπέρ κατά αποχές δεκτό εκα... ε, έλεγχος του 131 δεκτή 132 υπέρ κατά αποχές δεκτή 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 138 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 140 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 141 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 143 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 144 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος παρακαλώ στην 146. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση η Δεκτή. 15 προς 13. Δεκτή. 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος στην 147. Δεκτή. 148 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 153 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος παρακαλώ, άρχεται για την 153 πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 155 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 156 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. 156. Δεκτή. 160 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 158 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 161 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 162 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 166 καταπίπτει, αποσύρθηκε, 167 δεκτή, 168 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 169 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 191 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 172 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 193 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος στην 173 παρακαλώ. Δεκτή, 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 175 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 177 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 178 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ε, προφορική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 8 ε, υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Απορρίπτεται, απορρίπτεται η 11. 12 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 13, 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 16. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 17 υπέρ κατά ε, δεκτή, 18 υπέρ κατά 19 ε, υπέρ κατά δεκτή και η 18 είναι δεκτή. Πρέπει να ελέγξουμε τη 19 παρακαλώ, τη 19. Δεκτή, δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 εμπλουά υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ α καταπίπτει. 1 ε, ε, υπέρ κατά ε, αποχές δεκτή. Το 1 και το 2. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. φρίκι, λέει πρόεδρος. Ένα, αμπλουά. Λοιπόν, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, δεκτό. Τρία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Έξι, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Εφτά, υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε την εφτά, παρακαλώ. Δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 split vote. Πρώτο μέρος. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά... Α, την 23. Την 23 παρακαλώ. Δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος στις 24 παρακαλώ. Είπε έλξη ψηφοφορία. Δεκτή. 25. Όχι λέει. Όχι, 25. Α, ναι. 25. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές. 38 παρακαλώ έλεγχος. Έληξε δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε τη 43 Δεκτή. 44 υπέρ κατά εποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. 45. Δεκτή. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέραση ψηφοφορίας. 24, 25, 25 προς ε, μία ψήφο. Πολύ καλό αποτέλεσμα κυρία Χάνιμπολ, συγχαρητήρια. Στην We go a little bit faster now. We come to the local guard. Local guard? To local guard. You have to say something? Έχετε να πείτε κάτι για την επόμενη έκθεση Guard. Ένα σχόλιο. Η κατάσταση για την έκθεση αυτή δεν θα οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα ως προς τη φωνή της Πρόεδρου Υπάρχουν ορισμένες επεξηγήσεις ε, στο θέμα, αλλά η κυρία Παλιαδέλη θα επανέλθει σε αυτές. Είναι θέμα λεπτομέρειες όμως. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Δύο, Υπέρ, κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ τη δύο. Απορρίπτεται. προφορική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4. Λέει. Πάμε στο 4. Ναι, ναι. Ήμουνα, είχα δίκιο για μια φορά, λέει η πρόεδρος. <laughs> Το 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ κατά αποχές δεκτό, δεκτή. 7. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ κατά αποχές δεκτή, 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 13 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε τη 13 παρακαλώ. 13. Απορρίπτεται 13-14 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίστε 25 προς 2. Πάρα πολύ. Είμαστε ευτυχείς. Σας ευχαριστούμε κύριε Λόκεγκαρντ. Ήταν και αυτό ένα δύσκολο έργο. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Έχετε κάτι να πείτε κύριε Μιγκάλσκι. Όχι, ωραία, αρχίζουμε. Ένα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. The vote closed. Έληξε ψηφοφορία. δεκτεί Πάμε στη 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. δεκτεί 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. δεκτεί 5. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ στην 5. 5. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 25 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό, δεύτερο υπέρ κατά Απο, ε, αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά. Α, να ελέγξουμε την 26 παρακαλώ. Δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε τη 32. Δεκτή. 32 δεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 37. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 38. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 38. Λοιπόν, 18 προς 10. Δεκτή. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε συμβιβαστική 5. 15 προς 12 δεκτή. 45. Ε, 45. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση. της ψηφοφορίας. 26 προς 2. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Λόκεγκαρντ είπε πρόεδρο, αλλά τον κύριο Μιγκάλσκι θα εννοούσε. Λοιπόν, αυτέ οι φοβερέ τώρα ψηφοφορίε ε, ολοκληρώθηκαν. yeah. but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 Ε, θα ήθελα τώρα να επανέλθουμε στην επόμενη μας άσκηση που είναι μια ακρόση για ένα πολύ σημαντικό θέμα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση ευρωπαϊκή και η σημερινή κατάσταση. Αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ επίκαιρο γιατί έχουμε μία έκθεση για την Πολόνια, θα έχουμε επίσης και μία έκθεση για την ανακοίνωση της Κομισιόν και εάν θυμόσαστε μερικοί από εσάς Είχα παρουσιάσει τη γνωμοδότησή μου για την Πολόνια το 2008, η οποία ψηφίστηκε ε, στο, στην Ολομέλεια αφού συζητήθηκε στην Επιτροπή. Τώρα έχουμε προχωρήσει σε μερικά χρόνια και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Μερικά πράγματα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια αλλά ο βασικός στόχος της διαδικασίας της Μπολόνια ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος ε, της ανώτατης εκπαίδευσης, στην Ευρώπη το 2010 και η αύξηση της κινητικότητας στο επίπεδο αυτό. Και δεν μπορώ να πω ότι πραγματικά αυξήθηκε η κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε πολλούς τομείς πρέπει να πούμε, να ομολογήσουμε ότι πάρα πολλοί φοιτητέ δεν μπορούν πλέον να πάνε στο εξωτερικό ή σε μια άλλη χώρα, διότι το πρώτο τους πτυχίο είναι τόσο φορτωμένο που, που δεν προλαβαίνουν. Δεν, δεν μπορούν να επιβαρυνθούν περισσότερο. Και πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να έχουν την ευκαιρία να δούνε και να μάθουν κάτι διαφορετικό αντί να τους ε, φορτώνουν τόσα, τόσα πολλά μαθήματα και τόσο πολύ ύλη ε, στατικά ας πούμε σε ένα πανεπιστήμιο. Χαίρομαι που πήραμε μία ανακοίνωση από την Κομισιόν η οποία έχει ως στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι του, οι 20 με επικέντρωση βεβαίως στις θέσεις εργασίας, την εξέβρεση και διευκόλυνση στην πρόσβαση στην αγορά της εργασίας. Ε, είχαμε και το συνάλφο Καρλ Σμιτ, ο οποίος είναι πρόεδρος τώρα στην Ουγγαρία, ο οποίος είχε παρουσιάσει την έκθεση τότε ε, με θέμα πανεπιστήμια και οικονομία, οικονομικές εξελίξεις. Αυτό πάλι είναι εξαιρετικά επίκαιρο θέμα. Αυτό που με ευχαριστεί ιδιαίτερα είναι ότι η Κομισιόν πήρε την πρωτοβουλία και παρουσίασε στο Κοινοβούλιο μία ανακοίνωση η οποία, δεν, αυτή η διαδικασία δεν τηρήθηκε στην ε, διαδικασία της Μπολόνια. Η Κομισιόν έμεινε βουβή απλώς ε, ως παρατηρητής και τελικά διευθετήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο. Ε, βεβαίως η Κομισιόν χρησιμοποίησε τα θεσμικά μέσα, αλλά παρέκαμψε και ε, ε, στάθηκε σιωπηλή στην εξέλιξη της διαδικασίας της Μπολόνια. Τώρα η Κομισιόν ενεργεί πολύ σωστά, παρουσιάζει μια ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο και μαζί με την Κομισιόν, απαντώντας σε αυτή την ανακοίνωση, θα πιέσουμε το Συμβούλιο επιτέλους να κάνει κάτι ε, περισσότερα πράγματα σε αυτό τον τομέα. Τα λόγια δεν επαρκούν, πρέπει να πράξουμε, ε, πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αυτή την ακρόαση σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με εμπειρογνώμονες ε, από διαφορετικούς τομείς Έχουμε τον καθηγητή Τζούνιο Λουτσάτο, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Μπολόνια, τον κύριο Τζέριο Σάλιβαν, ο οποίος είναι επικεφαλής της ε, αρμόδιας αρχής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ιρλανδία, τον κύριο Μάρκο Μάτιλα από την Ακαδημία της Φιλανδίας και τον καθηγητή κύριο Φέντρινγκ, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας της, κοινωνίας των πολιτών, ε, της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών και υπεύθυνο για τη διαβίω εκπαίδευση. Καμία κυρία. Α, δεν έχουμε κυρία στο πάνελ. Ναι, αλλά ήρθατε, ανταποκριθήκαν οι καλεσμένοι μας στο πάνελ, στην πρόσκλησή μας και έχουμε και τον εισηγητή μαζί μας και είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να ασχοληθούμε εις βάσος με αυτό το θέμα. Κατά η πρώτη στην πρώτη φάση θα καλέσουμε να παρουσιάσουν την εισήγησή τους οι καλεσμένοι μας, οι εμπειρογνώμονες, 10 λεπτά ο καθένας. Χρόνο μιλίας, έχουμε εμείς το, στην Ορομέλεια μόνο τρία λεπτά. Το, αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Άρα πιστεύω ότι σε δέκα λεπτά που δίνουμε στους καλεσμένους μας θα έχουμε τη δυνατότητα να μας ε, κάνουν μια εμπεριστατωμένη εισήγηση για το θέμα αυτό. Εν συνεχεία θα έχουμε ερωταπαντήσεις. Ε, θα δώσουμε το λόγο και στην Κομισιόν ασφαλώς αν έχει κάτι να προσθέσει και η Πολωνική Προεδρία εάν εκπροσωπείτε εδώ. Α, ωραία, είσαστε εδώ κύριοι. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και κάτι άλλο, μια ένα τεχνικό ζήτημα. Σας θυμίζω ότι αυτή η συνεδρίαση παρουσιάζεται στο διαδίκτυο. Και, και τηλεοπτικά. Αυτό έχει άμεση σχέση με τη συμπεριφορά των συναδέλφων. Αν μπορείτε να μην κοιμηθείτε, ε, χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο σας εξ αριστερών ε, και επίσης πατήστε το μικρόφωνο να ανάψει το φωτάκι και όταν σταματήσετε να μιλάτε πατήστε πάλι για να κλείσει το φωτάκι. Λοιπόν, επίσης χαιρετίζω τον καθηγητή κύριο Μάτσινα, ο οποίος είναι υφυπουργός και τον κύριο Άντρες Κούκεβιτς Α, είναι διευθυντή του τμήματος του εκπαίδευση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεία και τον κύριο Άλαν Τούσον, μόλι ήρθε. Γενικός διευθυντή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ε, στην, ε, στο Εράσμο, στη Διεύθυνση Εράσμος. Και θα αρχίσω με τον κύριο Λουτσάτο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα να αναφέρω σύντομα κάποιες ε, ιδέες τις οποίες εξετάσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση των Υπουργών στην ε, Λουβέν Λανέβ. Κατά τη διάρκεια της οποίας ε, Προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε τα δέκα πρώτα χρόνια της διαδικασίας της Μπολόνιας, καθώς επίσης και την έναρξη της νέας αυτής δεκαετίας όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα ξεκίνησαν όμως με τη διαδικασία της Μπολόνια, πριν από δέκα χρόνια, όπως το γνωρίζετε. Στον ανακοινωθέν της συνεδρίασης της Υπουργικής στη Λουβέν Λανέβα, αναφερθήκαμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Αυτά θα ήθελα να αναφέρω εγώ τώρα και τα υπόλοιπα σημεία θα τα αναφέρουν οι υπόλοιποι ομιλητέ ε, στη συνέχεια τη ε, συνεδρίαση αυτή. Δεν θα αναφερθώ δηλαδή στην κινητικότητα και στη διαβίου μάθηση, ούτε στη σχέση που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμια εκπαίδευση και Ευρωπαϊκού χώρου έρευνα, γιατί αυτά είναι τα θέματα που θα αναπτύξουν οι επόμενοι ομιλητέ. Όσον αφορά λοιπόν το ανακοινοθέν τη ε, Λουβέν, Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι όσον αφορά την χρηματοδότηση υπάρχει μια σημαντική φράση. Στα πλαίσια της, ευθύνης, της, στα πλαίσια της δημόσιας ευθύνης δεσμευόμαστε για την δημόσια χρηματοδότηση. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση καθώς επίσης και μεγαλύτερη ανάπτυξη των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η φράση αυτή για τη χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα θυμάστε ότι είναι το ανακοινοθέν του Βερολίνου του 2003, το οποίο ανέφερε ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό και δημόσια ευθύνη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το αποδέχονται όλοι στον κόσμο. Ορισμένοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μία αγορά για την εκπαίδευση. Η βασική αρχή όμως της διαδικασίας της Μπολόνιας ήταν να καθοριστεί ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό και γι' αυτό το λόγο υπήρχε και αυτή η ρητή δήλωση. Έχουμε στη συνέχεια βέβαια και την ε, δημόσια, την κοινωνική με συγχωρείτε διάσταση, καθώς επίσης και την ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση, και αυτή την βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στην διαδικασία της Μπολόνιας. Δεν έχουμε καταφέρει όμως να πετύχουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα ακόμα βρισκόμαστε ακόμα αρκετά πίσω σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει όσον αφορά την κοινωνική διάσταση. Βλέπετε εδώ πέρα μια γραφική παράσταση που αν δούμε τα στοιχεία που έχουμε από πάνω προς τα κάτω, βλέπουμε ότι έχουμε πάνω στην πρώτη λίστα, στην πρώτη γραμμή με συγχωρείτε, φοιτητέ οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφίες, στην κάτω γραμμή τους φοιτητέ από τις χώρες εκείνες που δέχονται λιγότερες υποτροφίες. Βλέπετε επίσης τους φοιτητέ εκείνους οι οποίοι πληρώνουν δίδακτρα, αυτούς που δεν καταβάλουν δίδακτρα και βλέπετε επίσης τις ε, χώρες εκείνες όπου έχουμε περισσότερους φοιτητές, λιγότερους φοιτητές, τι χώρες εκείνες που έχουν περισσότερες υποτροφίες, λιγότερες υποτροφίες, καθώς επίσης και τις χώρες εκείνες όπου έχουμε περισσότερα δίδακτρα ή χαμηλότερα δίδακτρα. Βλέπετε επίσης σχετισμό ανάμεσα στις δύο αυτές μονάδες, σχέση δηλαδή ανάμεσα στους φοιτητές που λαμβάνουν υποτροφίες, σε σχέση με τα δίδακτρα τα οποία πρέπει να καταβληθούν σε κάθε χώρα. Δεν θα αναφερθώ, όπως σας είπα, στη διαβίου μάθηση, θα αναφερθώ στην απασχολησιμότητα. Σαφώς υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αυτή τη στιγμή λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αναλυφθούν οι απαραίτητε δράσεις προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα τα προπτυχιακά πτυχία, τα bachelor. Για, σε ορισμένες χώρες τα πτυχία αυτά αποτελούν κάτι το καινούριο, άλλες χώρες παρέχουν τα πτυχία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Θα ήθελα να σας πω ότι ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ο κύριος Βίνκλερ, είπε στην Βιέννη, όταν είχαμε μια επέτειο τότε για, την, για τα 10 χρόνια της διαδικασίας της Μπολόνιας, είπε λοιπόν ότι η απασχολησιμότητα των πτυχιούχων που έχουν μπάτσελόρ αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες των κρατών μελών ή θα πρέπει να αποτελεί μία από τις πιο βασικές προτεραιότητες. Ακόμα και η δημόσια διοίκηση και οι δημόσιες υπηρεσίες στα κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν πλήρω το πτυχίο αυτό, το πτυχίο bachelor. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια πολιτική για τη σωστή αξιολόγηση και αναγνώριση των πρώτων πτυχίων, των πτυχίων bachelor όλα αυτά τα σημεία τα οποία διατρέχω αυτή τη στιγμή αποτελούν ουσιαστικά τις ε, πρωταρχικές προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία και αποτελούν ουσιαστικά τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης του ε, Λέβεν. Βλέπετε εδώ πέρα επίσης κάποια εξίσου σημαντικά σημεία, κάτι το οποίο έφερα και στην αρχή της ε, παρουσίασής μου, το ότι δηλαδή δεν έχουν γίνει ακόμα σημαντικά πράγματα προκειμένου να καταφέρουμε να πείσουμε όλους τους καθηγητές στα πανεπιστήμια για αυτά τα οποία έχουμε θέσει εμείς ως βασικές αρχές στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο τα προγράμματα στα, σε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τις, σπουδε, σπουδές των φοιτητών και όχι τόσο στο, περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό των σπουδών, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξατομικευμένες δεξιότητες και τα ταλέντα που έχουν οι φοιτητές και ότι θα πρέπει να προωθηθούν οι δυνατότητες διαβίου μάθησης. Ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επίσης ε, δείκτε του Δουβλίνου, καθώς επίσης και άλλα συστήματα αξιολόγησης πανευρωπαϊκά και ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένε κατευθυντήριες γραμμές και συστήματα συγκριτικής αξιολόγησης. Θεωρητικά ισχύουν όλες αυτές οι αρχές, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτές από όλους τους καθηγητές και τους διδάσκοντες στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Πρέπει επίσης να Υπάρχουν σε πρακτικέ, οι οποίε ήταν γνωστέ από όλου του διδάσκοντε σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα πρέπει επίση να κάνουν περισσότερα τα πανεπιστήμια προκειμένου να καταφέρουν να καταρτήσουν καλύτερα τους δικούς τους διδάσκοντες όσον αφορά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Θα πρέπει δηλαδή οι καθηγητές πανεπιστήμια να γνωρίζουν πλέον τις νέες αυτές τεχνικές, καθώς επίσης και τις νέες μεθοδολογίες στη διδασκαλία, οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν πανευρωπαϊκά. Θα γίνει μια παρουσίαση για τη διαβίου μάθηση. Δεν έχω να πω κάτι αυτή τη στιγμή για την κινητικότητα. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, μια διαφάνεια η οποία δεν θέλει να εμφανιστεί στην οθόνη. Θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή για την ελαστικότητα, την ευελιξία στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα προγράμματα δασκαλίας. Και αυτό είναι εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο στα πλαίσια της κινητικότητας και της διαβίου μάθησης. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία να επικεντρώνονται στις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, αλλά αν είναι πάρα πολύ εξατομικευμένα τα, προβλήματα, τα, τα προγράμματα αυτά, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως τροχοπέδι στην κινητικότητα των φοιτητών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να, να μιλήσουμε και για συγκεκριμένα εργαλεία, όχι μόνο για δείκτες. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία. Καλύτερη οργάνωση των δεδομένων. Στο παρελθόν υπήρχε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της Μπολόνιας και είχαμε πει τότε ότι η αξιολόγηση αυτή δεν θα μπορούσε ποτέ να ολοκληρωθεί πλήρως ή δεν ήταν πλήρως ολοκληρωμένη ακριβώς επειδή δεν είχαμε τα απαραίτητα δεδομένα ή και τα δεδομένα που είχαμε δεν ήταν ομογενοποιημένα, δεν ήταν απόλυτα συγκρίσιμα. Πρέπει λοιπόν και αυτό να αποτελέσει ένα στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει προκειμένου να έχουμε μία ομογενοποιημένη γενική ομοιόμορφη οργάνωση των δεδομένων. Σε, κράτη, ορισμένα κράτη δεν είναι εύκολο να συλλεχθούν τα δεδομένα από τα πανεπιστήμια. Πάντως το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε πραγματικά την επόμενη δεκαετία να πετύχουμε αποτελέσματα μετρήσιμα και αξιολογήσιμα. Ένα ακόμα σημείο το οποίο θέλω να θίξω έχει να κάνει με διάφορα πολυδιάστατα εργαλεία για την διαφάνεια. Έχουμε, ξέρετε, τις ταξινομήσεις των πανεπιστημίων και των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πολλές φορές όμως οι ταξινομήσεις αυτές επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς και πτυχές. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση Όσον αφορά τη στάση των πανεπιστημίων στην ανάληψη δράσεων προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική διάσταση και πρόσβαση στην πανεπιστημία. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολυτομεακές πολυσχηδείς ταξινομήσεις και αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητα στα μέσα τα οποία διαθέτουμε για να αξιολογούμε όχι μόνο την έρευνα στα πανεπιστήμια, αλλά και άλλους στόχους και άλλες αποστολές των πανεπιστημίων. Έφτασα στο τέλος της παρουσίασής μου. Αυτό το οποίο θέλω ακόμα να πω είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα επαρκή συντονισμός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμέρους κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δύο διαφορετικά πλαίσια προσόντων. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, το οποίο ε, δημιουργήθηκε προκειμένου να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε και τη διαβίου μάθηση ως αναπόσπαστο στοιχείο, δεν συνάδει όμως με τη διαδικασία του Δουβλίνου που προβλέπεται για τα επίπεδα 6, 7 και 8 που ανταποκρίνεται δηλαδή στα, σημεία, στα πτυχία bachelor, master και διδακτορικό πτυχίο. Τα δύο συστήματα είναι συμβατά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Η συμβατότητα δεν αρκεί. Πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε κάποια πανεπιστήμια να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τα πτυχία τους σε ένα γενικευμένο σύστημα διαβίου μάθησης. Το να λειτουργούμε αυτή τη στιγμή με δύο παράλληλα συστήματα προφανώ δεν μα διευκολύνει. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμό. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας πω ότι απευθυνθήκατε και με αγγίξατε στην καρδιά. Ο κύριος Σάλιβαν έχει στη συνέχεια το λόγο που είναι υπεύθυνο για τα προγράμματα Εράσμους από πλευρά Ιλλανδίας. Έχετε το λόγο, κύριε Σάλιβαν. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ο αρχικός τίτλος ήταν «Μαθήματα από την Ιρλανδία», αλλά θα μπορούσα να σας μιλήσω για την δική μας εμπειρία και πήρα σε σχέση με την ανώτατη εκπαίδευση. Για να μιλήσω μέσα σε εθνικά πλαίσια θα ήθελα να πω ότι ιστορικά είχαμε μεγάλη πείρα σε αυτό το τομέα, γιατί ιστορικά δεν είχαμε τόσους πόρους και άλλες χώρες είχαν ε, μεγαλύτερη βιομηχανία, καλύτερη οικονομία και οικονομικές δυνατότητες, γι' αυτό εμείς σταθήκαμε στην εκπαίδευση. Και βεβαίως η κινητικότητα είναι αναπόσπαστο μέρος, διότι έπρεπε να ανταποκριθούν, να μεταβούν αλλού. Τώρα η κινητικότητα είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και οι Ιρλανδοί φοιτητές έχουν αγκαλιάσει αυτή την έννοια. Θα ήθελα να σας δείξω μία διαφάνεια για να δείτε πώς η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκπαίδευση έφτασε σε μια κατακόρυφη ανάπτυξη και μετά έπεσε λίγο λόγω δημογραφικών αλλαγών, αλλά αυξήθηκε ενέου, εκ νέου πρόσφατα. Και αυτό σήμαινε ότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου το 65% των 17χρονων πηγαίνουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι το υψηλότερο ποσοστό ανά τον κόσμο. Και θα ήθελα να πω ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ε, δρούν διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα, γιατί ανταποκρίνονται στις τοπικές πολιτισμικές και ιστορικές ανάγκες. Όταν μιλάμε λοιπόν για ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε σχέση με την ιστορική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι χώρες και η Ιρλανδία δεν αποτελεί εξαίρεση διότι έχει συμμετοχή στα ΑΕΗ πολύ μεγαλύτερη από τα άλλα κράτη-μέλη και στο τομέα της κινητικότητας υπήρχε διαφορετική εξέλιξη ανάλογα με τις ανάγκες του δυτικού κόσμου. Μιλάμε για τις αγγλόφωνες χώρες όπου βλέπουμε ότι οι Ιρλανδοί μεταβαίνουν στις ΗΠΑ και στην υπηρετική Ευρώπη. Στο 18ο αιώνα πολλοί Ιρλανδοί πολλά εκατομμύρια πήγαν στην Ευρώπη και πήγαν βεβαίως και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Um, Όταν η Ιρλανδία συμμετείχε στη διαδικασία της Μπολόνια, το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα είχε, μάλλον ε, ακολουθούσε τη διαδικασία της Μπολόνια. Είχαμε δηλαδή ένα εκπαιδευτικό σύστημα τριών κύκλων. Και σύμφωνα με την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε και την κοινωνική διάσταση. Η ανώτατη εκπαίδευση διανύει μια περίοδο αλλαγών. Ίσως προχωρήσαμε περισσότερο σε σχέση με τους στόχους ε, της Μπολόνια και δεν υπήρχαν τόσο τραυματικές εμπειρίες στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα γιατί το σύστημά μας συνάδει με αυτό το πρότυπο που προτείνει η διαδικασία της ε, Μπολόνια. Και οι προτεραιότητες ε, της ανώτατης εκπαίδευσης της Μπολόνια ήταν σε συμμετρία με το εθνικό μας σύστημα. Από στην αρχή είχαμε ένα σύστημα χαρτογράφησης που, όπου συμμετείχαν όλες, ε, όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όπως ίσχυε στη διαδικασία της Μπολόνια και στην Ευρωπαϊκή Διαδικασία Προσόντων. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπου η Ιρλανδική εμπειρία μας βοήθησε γιατί υπήρχε κυβερνητική υποστήριξη για όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες. Και είχαμε και διάφορους ε, φορείς, όπως τον Εθνικό Φορέα Προσόντων, καθώς και έναν Εθνικό Φορέα Πρόσβαση στην ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου λαμβάνουμε υπόψη τις εθνοτικές μειονότητες, τους ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας και ούτω καθεξής. Άρα είχαμε επιμέρους στοχοθετήσεις και ήθελα να τονίσω ότι υπήρχε πάντα εθνική υποστήριξη στην συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση και βεβαίως με βάση το Εράσμους από το 1998 συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα κινητικότητας που είναι το υψηλότερο επίπεδο κινητικότητας. Υπάρχουν και άλλοι φορείς ποιοτικού ελέγχου όπου συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και υπήρχε και συμμετοχή, ευρύτατη συμμετοχή του δημόσιου τομέα. Αυτό είναι αρκετά θετικό για μία τόσο μικρή χώρα. Αυτή η διαδικασία λοιπόν οδήγησε σε μία ευελιξία. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις εθνικές και τις διεθνείς ανάγκες. Άρα σε αυτή τη ε, διαδικασία της Μπολόνια, σε αυτή την περίοδο, υπήρχε, ε, δόθηκε μια μεγάλη όθηση για ε, μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα για την κινητικότητα των φοιτητών μέσα στα πλαίσια και της ε, διαδικασίας για το 2020. Και το πρόγραμμα Έρασμος ε, ήταν πολύ σημαντικό γιατί 250.000 φοιτητές συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και περίπου 3 εκατομμύρια θα έχουν φτάσει σε αυτό το στόχο μέχρι το 2013. Τα τελευταία πέντε λοιπόν χρόνια αυξήθηκε η συμμετοχή στο πρόγραμμα Έρασμος και ο Εθνικός Φορέας Εκπαίδευσης έδωσε και μία μεγάλη όθηση Και θα ήθελα να πω ότι αυτό βοήθησε διότι ενθάρρυνε τους φοιτητέ να έχουν ένα σχετικό πλεονέκτημα όταν αναζητούν μία εργασία. Και νομίζω ότι για να προωθήσουμε αυτές τις δυνατότητες, αυτή την υψηλότερη κινητικότητα, πιστεύω ότι τα Υπουργεία Παιδείας θα πρέπει να τονίζουν αυτή τη δυνατότητα του σχετικού πλεονεκτήματος, το οποίο δεν γίνεται πάντα κατανοητό ούτε από τους εργοδότες. Θα φτάσουμε από 2,5 σε 3.000 σε αυτή την πρώτη φάση της διαβίου μάθησης. Ως προς τα πρότυπα κινητικότητας, βλέπουμε ότι αυξάνεται η κινητικότητα, αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος η κινητικότητα να λάβει επιτόπιο χαρακτήρα. Και η δική μας πείρα δείχνει ότι τα δύο τρίτα των φοιτητών πάνε σε δύο-τρεις χώρες χώρες που, όπου η γλώσσα των οποίων μαθαίνεται κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και γι' αυτό υπάρχουν προσκόμματα πολλές φορές και γι' αυτό αναζητούν χώρες όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά. Υπάρχει μία πολύ μικρή αλλαγή και γι' αυτό βλέπουμε ε, ότι οι περισσότεροι μεταβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα 65%. Βεβαίως και στις ανθρωπιστικές σπουδές και στις νομικές σπουδές υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δεν υπάρχει δραστηριότητα σε τομείς όπως των ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων ή μηχανικών. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι το ανώτατο ε, σύστημα, το ανώτατο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι ύψης της σημασίας ε, γιατί πιστεύουμε ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια και της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Έχει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και για την ποιότητα των γνώσεων και μας ενδιαφέρουν και νέες δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας έτσι ώστε να είναι καλύτερα απασχολήσιμοι οι φοιτητέ μας στο μέλλον. Και αυτό, σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η κινητικότητα. Θα πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα στο γλωσσικό, προς το γλωσσικό μας καθεστώς, γνωρίζοντας περισσότερες ε, ε, ε γλώσσες και υπάρχουν μεγαλύτερες συνέργειες και με άλλους φορείς και ιδρύματα όπως το Marie Curie και άλλα. Θα ήθελα να πω όμως ότι σε επίπεδο κυβέρνησης υπάρχει η θέληση να γίνει αυτό. Και ο μιλητής χαιρέτησε στα γκέιλικ, στα κελτικά. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο μίλησατε για ε, studies placements. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Erasmus, έχουμε συμμετοχή σε 4.000 πανεπιστήμια, μπορούν δηλαδή να μεταβούν σε ένα άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από 3 μέχρι 12 μήνες. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Στη δεύτερη μπορούν κατά την ίδια διάρκεια να παρευρεθούν σε μία επιχείρηση και να εργαστούν αντί να, ε, αντί να σπουδάσουν. Δηλαδή σαν να πρόκειται ένα είδος στάζ σε μία επιχείρηση. Ναι, σας ευχαριστώ γιατί δεν το κατανόησα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στον επόμενο μιλητή, τον καθηγητή Μάρκου Μάτιλα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ μεγάλη ευχαρίστηση που μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω την παρουσίασή μου αυτή για τις καλύτερες συνέργειες ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 που ουσιαστικά στοχεύουν σε μία ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται στην γνώση και την καινοτομία. Στον πυρήνα της στρατηγικής αυτής βρίσκεται το περίφημο τρίγωνο της γνώσης, το οποίο περιλαμβάνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε αυξανόμενη συνεργασία ανάμεσα στα τρία αυτά σημεία, εκπαίδευση, έρευνα και κοινοτομία. Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας τώρα. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται για περίπου 10 χρόνια. Με την συνθήκη της Λισαβόνας έχει πλέον νομική βάση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική αλλαγή. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας ουσιαστικά σημαίνει καλύτερη χρήση του ανθρώπινου και οικονομικού δυναμικού που υπάρχει στην Ευρώπη για την έρευνα. Ο βασικός στόχος είναι να καταφέρουμε να καταρρύψουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στη διασνοριακή έρευνα και κατά αυτόν τον τρόπο να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Υπάρχουν πολλές αλληλοσυνδέσεις και συνέργειες ανάμεσα στις δύο, στους δύο αυτούς χώρους. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι σημαντικοί φορεί σε κάθε περίπτωση. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τρετοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας ουσιαστικά έχουν κοινούς στόχους. Έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και να καταστήσουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα πιο δημοφιλή. Και σίγουρα μπορούν να συμβάλλουν και οι δύο αυτοί χώροι στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα μας επιτρέψει να αποκριθούμε στις πολύ μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Προκειμένου να πετύχουμε το στόχο αυτό, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας υποστηρίζει την έρευνα εχμής, η οποία έρευνα μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην αύξηση της ποιότητας των ονότατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης. Η κατάταξη των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων στι παγκόσμιε κατατάξει ανώτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ουσιαστικά έχει να κάνει με την ποιότητα τη έρευνα πάρα πολλέ φορέ. Έχουμε ε, διάφορους φορείς χρηματοδότησης τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η Ακαδημία της Φιλανδίας, την οποία εκπροσωπώ. Τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να προσφέρουν μια σημαντική, ένα σημαντικό επίπεδο εκπαίδευσης παγκοσμίως, αν δεν είναι σε θέση να παρέχουν και μια ποιοτική έρευνα. Ένας άλλος κοινός στόχος είναι η μεταφορά γνώσης ανάμεσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την κοινωνία. Ο στόχος αυτός είναι κοινό και για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα και για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε όμω εδώ νέε δομέ προκειμένου τα τελευταία πορίσματα της ε, έρευνας εχμής να γίνονται πιο εύκολα διαθέσιμα στους πολιτικούς ηθήνοντες, αυτούς που χαράσουν πολιτική στα κράτη-μέλη. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα πορίσματα της έρευνας σε διάφορους φορείς της κοινωνίας και σε διάφορες επιχειρήσεις. Καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Τα κέντρα αυτά τα οποία έχουμε στη Φιλανδία συνδέονται και με τα συστήματα διδακτορικών προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν στην πανεπιστήμια μας. Ένα άλλο θετικό παράδειγμα της επιτυχίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας είναι η έννοια των Ευρωπαϊκών Κέντρων Τεχνολογίας και Κοινοτομίας, έννοια η οποία άρχισε να ισχύει από το 2008. Τα ENT λοιπόν αυτά δημιουργούν πράγματι ένα σύνδεσμο ανάμεσα στην έρευνα και την καινοτομία που παράγεται στα πανεπιστήμια και συμβάλλουν πάρα πολύ στην διάχυση της γνώσης. Παρέχουν διάφορα προγράμματα μεταπτυχιακά και ουσιαστικά συμβάλλουν στο να χρησιμοποιηθούν τα πορίσματα της έρευνας από τις επιχειρήσεις και προωθείται μια πολυτομιακή κινητικότητα καθώς επίσης και αύξηση της απασχολησιμότητας στον ιδιωτικό τομέα. Ένα από τα δυνατά σημεία των κέντρων αυτών είναι το ότι συμβάλλουν πάρα πολύ στην προώθηση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται στην τελευταία έρευνα που παράγουν τα πανεπιστήμια. Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες. Σε τελευταία ανάλυση, τα πανεπιστήμια δραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να δημιουργούν καινοτομία η οποία βασίζεται στην έρευνα. Νομίζω ότι μόνο οι καινοτομίε αυτέ που βασίζονται στην έρευνα μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν καλύτερε θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκό χώρο έρευνα και ο Ευρωπαϊκό χώρο Τριτοβάθμιση εκπαίδευση έχουν ε, κάποιες ακόμα κοινέ προτεραιότητες όσον αφορά τα προγράμματα εκπαίδευσης για τα διδακτορικά. Η διδακτορική εκπαίδευση θα πρέπει καταρχάς να γίνει πιο ελκυστική για τους νέους ταλαντούχους, υποψήφιους φοιτητές και τα διδακτορικά προγράμματα μπορούν να στεφθούν με επιτυχία αν τελικά οι φοιτητέ μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν σε μια έρευνα ανώτατης ποιότητας και να συμμετέχουν σε πραγματικές ερευνητικέ δράσει. Προκειμένου να καταρτήσουμε καλύτερα τους φοιτητές σε επίπεδο post-doc, θα πρέπει οι φοιτητές αυτές να είναι σε θέση να καταλάβουν τα τελευταία πορίσματα της πανεπιστημιακής έρευνας. Γι' αυτό το λόγο με σαφώς υπέρ των νέων αυτών αρχών της καινοτόμου κατάρτισης σε δακτορικά προγράμματα. Επίσης, η κινητικότητα σε δακτορικά προγράμματα ανάμεσα σε ε, ιδρύματα δημόσια διοίκηση, επιχειρήσει και πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι ένα καταπληκτικό τρόπος προκειμένου οι νέοι αυτοί να καταφέρουν ε, να βελτιώσουν τις δεξιότητέ τους. Η διατομιακή αυτή κινητικότητα επίσης είναι πολύ σημαντική για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για την πρόθεση της καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να χαιρετήσω τη νέα το νέο πολυτομιακό πλαίσιο για την πρόθεση των ε, της επαγγελματικής τεδρομίας στην Ευρώπη. Η κινητικότητα αυτή στα διδακτορικά προγράμματα παρέχει επίσης και μια εγγύηση για την ποιότητα. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλά εμπόδια για την κινητικότητα, όπως ακούσαμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε ακόμα τις απαραίτητες δομές προκειμένου να προωθήσουμε την κινητικότητα. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις διασυνοριακές συνεργασίες ανάμεσα στα διδακτορικά προγράμματα, ιδίως όσον αφορά το τομέα της έρευνας και θα πρέπει να καταρρύψουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν σε διάφορες κοινέ προσπάθειες κοινή έρευνας. Θα πρέπει να δημιουργηθούν κοινά προγράμματα διδακτορικών και όσον αφορά την εκπαίδευση, έχουμε το πρόγραμμα Erasmus Mundus, το οποίο αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για τέτοια κοινά προγράμματα διδακτορικών. Δυστυχώς όμως είναι λίγα τα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν στο Erasmus Mundus. Όσον αφορά την έρευνα έχουμε τις δράσεις Marie Curie, οι οποίες όντως έχουν συμβάλει στο να προωθηθεί η διεθνής κινητικότητα των ερευνητών και υπάρχει πλέον και μεγαλύτερη διασύνδεση με τον τομέα των επιχειρήσεων στα πλαίσια των δράσεων Marie Curie. Θα πρέπει πάντως να προωθηθούν τα υφιστάμενα προγράμματα κινητικότητας τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την έρευνα. Ένα παράδειγμα θετικής συνέργειας ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην έρευνα είναι το κοινό πρόγραμμα έρευνας και κοινοτομίας της Βαλτικής, που ανήκει στα προγράμματα του άρθρου 185. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής έχει ως στόχο να συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των προγραμμάτων και των ε, ηθήνων των πολιτικής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρικοδοτημένο με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί στα πλαίσια της, εκπαίδευση εκπαίδευσης και της έρευνας. Προβλέπονται επίσης προγράμματα κατάρτισης και κινητικότητας στα πλαίσια της περιφέρειας της Βαλτικής. Είναι ένα θετικό λοιπόν παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει περισσότερο σε νέα προγράμματα διδακτορικών, σε νέα προγράμματα έρευνας, τα οποία θα προωθήσουν στη συνέχεια και κάποια πιο προηγμένα προγράμματα καινοτομίας. Κυρίε και κύριοι, θεωρώ ότι ο Ευρωπαϊκό Χώρο Τροβάτμια Εκπαίδευση και ο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα είναι δύο έννοιε αλληλένδετε, οι οποίε αλλοϊποστηρίζονται. Χρειαζόμαστε όμω περισσότερε συνέργειε από αυτέ που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμή. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή τη όλη διαδικασία. Υπάρχουν τουλάχιστον έξι κοινά σημεία διεπαφή των δύο αυτών χώρων, αλλά υφίστανται ακόμη εμπόδια στην πλήρη υλοποίηση τη κοινή πρόθεση των δύο αυτών χώρων. Πιστεύω ότι τα εφιστάμενα εμπόδια θα πρέπει να ξεπεραστούν το συντομότερο δυνατό. ευχαριστώ. κύριε καθηγήτα και επόμενο ομιλητή είναι ο Καθηγητή, κύριος Μισελ Φέτρι. Έχετε το λόγο. Θα σας προβάλλω ε, το θέμα υπό μία διαφορετική οπτική γωνία από τους τρεις προλαλήσαντες, προσπαθώντας να διευρύνω τη σκέψη μας την πλατφόρμα σκέψης μας, διότι πολλές φορές η προσέγγιση μας αφορά τους νέους φοιτητές. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι στα πανεπιστήμια μας υπάρχει ένα διαφοροποιημένο κοινό που απαρτίζεται από ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Γι' αυτό θα πρέπει να διευρύνουμε τη βάση συλλογιστικής μας και αυτό θα ήταν σωστό και για τους ε, παρευρισκόμενους φοιτές και αποτελεί και μία αναγκαιότητα. Το άλλο στοιχείο αφορά την διαβίου μάθηση, lifelong learning, γιατί νομίζω ότι αν κάνουμε μία προβολή εδώ στην αίθουσα, ο καθένας θα είχε τη δική του οπτική γωνία, το δικό του ορισμό ως προς τη διαβίου μάθηση. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτές τις έννοιες. Αυτό που έχει σημασία σήμερα για τα πανεπιστήμια και για τις οικονομίες μας είναι να λάβουμε υπόψη ότι η διαβίου μάθηση δεν είναι επιλογή, δεν είναι μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά μια οικονομική αναγκαιότητα. Και νομίζω ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των κοινωνιών μας βασίζεται όχι μόνο στην επικαιροποίηση γνώσεων και προσόντων, αλλά στην επιτάχυνση της κίνησης αυτής, δηλαδή της τεχνογνωσίας και της εφαρμογής τεχνικών γνώσεων. Και σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαβίου μάθηση γιατί το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια είναι η παραγωγή ε, γνώσεων, είναι ο παραγωγός γνώσεων, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όταν ένα 50% ενός ηλικιακού φάσματος φτάνει στην ανώτατη εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο ασχολείται με αυτούς και θα έπρεπε με αυτή την, το ηλικιακό φάσμα και θα έπρεπε να ασχολείται και με το, το ηλικιακό φάσμα το οποίο άπτεται του ε, σκέλους της διαβίου μάθησης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ενιαία λοιπόν σταδιοδρομία, αλλά για ένα σύνολο σταδιοδρομιών για όλους. Γι' αυτό τα εθνικά μας ιδρύματα θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την αναπτυξιακή δυνατότητα σταδιοδρομιών στο διηνεκές. Άρα μιλάμε για διαχείριση αυτών των interface, των σημείων διεπαφής δηλαδή των διαφόρων σταδιοδρομιών και να δούμε πώς μπορούν να συμμετάσχουν και στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό, επιλέγοντας ένα επάγγελμα. Σήμερα τα πανεπιστήμια συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα, το εξελικτικό σχήμα, διότι πολλοί ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας επανέρχονται στα πανεπιστήμια. όπου έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές μονάδες και τα πανεπιστήμια δεν θεωρούν ότι αυτό είναι το επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους, δηλαδή δεν υπάρχει μία πραγματική στρατηγική όλα, όλοι αυτοί οι φοιτητέ μεγαλύτερης ηλικίας εντάσσονται σε περιφερειακά σχήματα των πανεπιστήμιων. Θα έπρεπε λοιπόν τα πανεπιστήμια να παρέχουν μακροχρόνια σχήματα μια μακροχρόνια βάση εκπαίδευσης έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να επανέλθουν οποιαδήποτε στιγμή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας για να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες. Δηλαδή να έχουμε να κάνουμε με άλλα σχήματα εκμάθησης για επικαιροποίηση γνώσεων και για μια νέα γνωστική βάση. Θα πρέπει λοιπόν να το εξασφαλίσουμε αυτό στους φοιτητές μας, δηλαδή να υπάρχει μία συνέχεια γνωστικών σχημάτων και μία ευελιξία έτσι ώστε να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να ανταποκριθούν όταν επανεγγράφονται φοιτητές, πρώην φοιτητές μας αργότερα, σε κάποια άλλη φάση της ζωής τους. Ε, βεβαίως είχαμε και πολλές πρόσφατες ε, πρωτοβουλίες. Είχαμε την ανακοίνωση των Υπουργών στο Λέβεν, στη Λουβέν, τον Απρίλιο του 2009 και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε άλλα σχήματα της ε, διαβίου μάθησης που είναι ένα σχήμα της Μπολόνια πέρα από το 2010, καθώς και οι προκλήσεις ε, με βάση το 2020, αλλά έχει μεγάλη σημασία το να περάσουμε από τη ρητορία στην πράξη. Τα πανεπιστήμια ανακοινώνουν τις στρατηγικές τους, μιλάνε για 35% το 2003 και 39% μέχρι το 2009 ε, επίπεδα συμμετοχής στη διαβίου μάθηση μέσα στα πλαίσια αυτής της διαβίου κατάρτισης μπορώ να πω. Πολλά προγράμματα αναπτύχθηκαν μέσα στα πλαίσια των ε, ευρωπαϊκών δικτύων ανώτατης εκπαίδευσης και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι συμβαίνει σήμερα στην ανώτατη εκπαίδευση. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι έχουμε τρία επίπεδα ε, στρατηγικής μέσα στα πλαίσια της ε, διαβίου μάθησης. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια που θεωρούν ότι πρόκειται για ένα στάδιο προσαρμογής, δηλαδή μιλούν για εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες δεν εντάσσονται στις πανεπιστημιακές δομές, ενώ παράλληλα μιλάμε για διαβίου μάθηση η οποία εντάσσεται στον πανεπιστημιακό ιστό. Έχουμε να κάνουμε με μια πολύ χαμηλή όμως ποσοστή αναλογία σε επίπεδο πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε σε ένα επίπεδο οργάνωσης όπου να έχουμε την αρχική κατάρτιση και στη συνέχεια την διαβίου κατάρτιση ή εκμάθηση. Έτσι θα πρέπει να έχει η δομή του Πανεπιστημίου. Για να έχει και ένα σκέλος, ένα ενταγμένο σκέλος που να αφορά τη διαβίου μάθηση, όπου να παρέχει νέες υπηρεσίες, υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν στις, ε, σε θετικές σταδιοδρομίες, στην εξέλιξη σταδιοδρομίας με βάση το γνωστικό και εκτιμένο, το μέχρι τούδε γνωστικό και εκτιμένο. Θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε και ένα τρίτο στάδιο, γιατί δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στην Ευρώπη που να έχει φτάσει αυτό, σε αυτό το στάδιο, να μιλήσουμε ε, δηλαδή για ένα πανεπιστήμιο όπου η διαβίου μάθηση εντάσσεται σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο, σε πολιτισμικά δεδομένα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε βεβαίως ότι αυτή η ενιολογική βάση ε, που αφορά τη διαβίου μάθηση μπορεί να οδηγήσει και σε έρευνες αριστείνδυν. Τρεις, πέντε είναι οι στόχοι. Καταρχήν θα πρέπει να διαρθρώσουμε πολύ καλά τις, ε, τα τρία στάδια, την αρχική ε, γνώση και την συνεχόμενη εκπαίδευση και έρευνα, να, μας, να λάβουμε ως επίκεντρο αυτόν ο οποίος είναι ο διαβίου φοιτητής μας ο learner και επίσης να λάβουμε υπόψη όλο το προσωπικό και όχι ε, μόνο τους διδάσκοντες. Και αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές μας θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα για τη διαβίου μάθηση. Και επίσης η κοινωνία θα πρέπει να είναι κοινωνός αυτής της ενιολογικής βάσης, αυτού του ενιολογικού σκεπτικού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φετρή. Και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ποιος θέλει παρακαλώ να λάβει το λόγο. Ε, σύντομα παρακαλώ και επί της ουσίας. Η κυρία Παλιαδέλη. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας για να μιλήσει στην, στα ελληνικά. Ε, κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι είμαι παρούσα σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, σε μια περίοδο μάλιστα που στην Ελλάδα ένας καινούριος νόμος ε, που έγινε αποδεκτός με μεγάλη πλειοψηφία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ε, αμφισβητείται από τους πανεπιστημιακούς και τους φοιτητές. Ε, περνάμε μια, ένα κομμάτι μιας κρίσης που έχει και στο Πανεπιστήμιο τις επιπτώσεις της. Θα πω κάτι που ίσως οι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή το έχουν ξανακούσει να λέω, αλλά είναι μια ερώτηση η οποία με απασχολεί συνεχώς. Βλέπουμε τα πανεπιστήμια της Ευρώπης ε, να ακολουθούν τα αγγλοσαξονικά πρότυπα θα έλεγα. Ε, αναρωτιέμαι αν ένα μέρος αυτής της ευρωπαϊκής κρίσης ε, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν έχει σχέση πιθανόν με αυτό το μοντέλο. Ε, τελευταία έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο για την ε, χρησιμότητα των ανθρωπιστικών σπουδών στην, στη δημοκρατία, τη συμβολή των ανθρωπιστικών σπουδών στη δημοκρατία. Η ερώτηση μου λοιπόν προς όλους τους ομιλήσαντες αφορά Πρώτον, την ανάγκη, ε, αν, έχει ε, επιληφθεί, ε, επιληφθούν αυτές, αυτοί οι δύο χώροι για την ανώτατη εκπαίδευση και για, την ευρωπαϊκή, για τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, το European Ranking. Έχουμε ανάγκη να ενός μιας μεθόδου μέτρησης των επιδόσεων των πανεπιστημίων βασισμένων σε ευρωπαϊκά κριτήρια. Όχι σε αυτά που καμιά φορά αμφισβητούμε και τα οποία επηρεάζουν και τον τρόπο σπουδών και τα κουρίκουλα κλπ. Ε, νομίζω ότι είναι απαραίτητο ένα ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγηση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Σε μιας αξιολόγηση που θα λαμβάνει υπόψη και την πολιτιστική εκδοχή των σπουδών ενώ τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Ε, θα καταλήξω ε, με μία ερώτηση προς όλους που έχουν μιλήσει πώς εννοούν την ε, καινοτομία σε χώρους που δεν είναι αναγκαστικά των θετικών επιστημών. Τι μπορούν να κάνουν όσοι υπηρετούν τις λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, προκειμένου να συμμετάσχουν ή να αξιολογηθούν από ε, ε, με, με κριτήριο την καινοτομία. Ένα είναι αυτό. Αυτή η ερώτηση για τη γενοτομία αφορά και στην έρευνα. Πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να αξιολογηθούν ε, επιστήμες χώροι ε, επιστημονικοί οι οποίοι ε, ανήκουν, ε, οι δεν εντάσσονται σε αυτό που ονομάζουμε ε, science. Πιστεύω ότι ορισμένες ανθρωπιστικές επιστήμες, ανάμεσα σε αυτές και αυτή που υπηρετώ εγώ τα πολλά χρόνια η αρχαιολογία είναι science, είναι μια επιστήμη, δεν είναι μόνο ανθρωπιστικές σπουδές. Θέλω να πω ότι μήπως οι όροι αυτοί, innovation και research αποθαρρύνουν όσους ασχολούνται με επιστήμες οι οποίες δεν υπάρχονται σε αυτόν τον κύκλο που, ε, αφορά, ε, ε, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ευρωπαϊκές σπουδές. Εκτιμώ ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και εδώ ε, ο χώρος ε, έρευνας είναι πολύ σημαντικός να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις επιστήμες και σε ό,τι αφορά την ε, καινοτομία και σε ό,τι αφορά την έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ γιατί θέσατε πολύ σωστά, σε σωστές βάσεις ε, τη συζήτησή μας, ε, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά παρουσίασε μία ανακοίνωση επί του θέματος. Και μετά από την έκθεση ΠΑΚ το 2009, χρειάζεται επικαιροποίηση της αξιολόγησης για να δούμε τι συμβαίνει στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια και στον, ε, στα ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βεβαίως, διανύουμε μία περίοδο μεγάλης οικονομικής ε, κρίσης, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη στην καθημερινή μας εργασία. Και τα πανεπιστήμια δεν ε, μπορούν να αποτελέσουν από μονομένες οντότητες μεταξύ τους. Θα πρέπει να κινούνται παράλληλα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες υπό τις οποίες η ολοκλήρωση να αφορά και, την, ε, και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ε, ιδρύματα και την έρευνα. Να μιλάμε για ανώτατα, ε, ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευρωπαϊκή έρευνα. Και θα πρέπει να προωθήσουμε νέα στοιχεία να μιλάμε για single market, για ενιαία αγορά, η οποία όμως δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρχει ενιαίος χώρος εργασίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε υψηλό εκπαιδευτικό, υψηλό επίπεδο παιδείας, έτσι ώστε ο κάτοχος ενός τίτλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος να ισχύσει και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα, διότι η διαδικασία της Μπολόνια και η ανώτατη εκπαίδευση είναι έννοιες που έχουν επινοηθεί αλλά δεν έχουν τύχει υποστήριξης αυτή την περίοδο. Δηλαδή είναι έννοιες κενές περιεχομένου εμπολής. Και γι' αυτό αυτό το νόημα έχει και η ανακοίνωση. Δηλαδή κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα και κάθε κράτος θα πρέπει να προχωρήσει και να λάβει υποστηρικτικά μέτρα υπέρ της διαδικασίας, τη της Μπολόνια και τα πανεπιστήμια να συγκλίνουν, να βρεθούν σε ένα επίπεδο σύγκλησης μεταξύ τους και θα πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους στα πλαίσια της διαδικασίας. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει bachelor, τι σημαίνει, ίσως είναι άλλο ε, για τις αγγλοσαξονικές χώρες, δηλαδή αφορά έναν τριετή κύκλο σπουδών που έχει ε, μία επαγγελματική διέξοδο. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο απασχολησιμότητας, employability. Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε σε μία από αξιολόγηση, διότι η αμοιβαία αναγνώριση αφορά και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εάν σε μία χώρα πάει ένας πτυχιούχος ιατρικής, ας πούμε ένας Ιταλός στη Γαλλία και οι Γάλλοι δεν θεωρήσουν καλό το επίπεδο σπουδών, δεν θα επιτρέψουν σε αυτό το γιατρό να ασκήσει το επάγγελμα. Άρα υπάρχει και θέμα αμοιβαία ε, ε, εμπιστοσύνης. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη ε, quality assurance. Και θα ήθελα να πω ότι τα κράτη, τα πανεπιστήμια, οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε η διαδικασία της ε, Μπολόνια να αλλάξει άρδιν τις δομές του Πανεπιστημίου. Γιατί από τεχνικής υφής δεν μιλήσαμε για τη διαδικασία της Μπολόνια, μιλήσαμε για στοχοθέτηση των πανεπιστημίων. αλλά η διαδικασία αφορά την ίδια την φύση των πανεπιστημίων και αυτό δεν μας απασχόλησε. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μπερλίνγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες που μίλησαν και τον κύριο Σάλιβαν οι εισηγήσει ήταν ενδιαφέρουσε, αλλά δεν αναφέρθηκαν στην ουσία του προβλήματος στην οποία αναφερθήκατε εσείς. Όσον αφορά δηλαδή την κινητικότητα. Η κινητικότητα ε, φοιτητών, μαθητών, ακαδημαϊκών, καθηγητών και ειδικά μια κινητικότητα προσαρμοσμένη στην απασχολησιμότητα και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πρέπει να αυξήσουμε την κινητικότητα αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Έχω ε, μερικές παρατηρήσεις και θέλω να ρωτήσω τους ομιλητές αν πιστεύουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Στο να ευθυγραμμιστούν τα, οι με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, έχουν προσταρμοστεί, έχουν εξυγχρονιστεί οι σπουδές, το περιεχόμενο σπουδών, ανάλογα με τις ανάγκες των ε, αγορών εργασίας. Δεύτερον, ένα σημείο το οποίο αναφέρθηκε. Η κατάσταση ε, των στέλεχων, των ανθρώπων, που δουλεύουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι καθηγητέ, δηλαδή το ακαδημαϊκό προσωπικό, εξαρτάται από τον αριθμό των μονογραφιών και των δημοσιεύσεων που έχουν κάνει. Ε, είναι σωστό αυτό. Υπάρχει ένα άλλο ή ένα καλύτερο σύστημα αξιολόγησης. Επίσης πρέπει ε, να δούμε εάν ε, τα προσόντα των καθηγητών ανταποκρίνονται στα προσόντα που λαμβάνουν οι φοιτητέ τους όταν αποφοιτήσουν. Δηλαδή, ο καθηγητή με χι τίτλους έχει δώσει τα χι προσόντα συν παραπάνω στους φοιτητέ που εκπαίδευσε. Ε, πολλοί φοιτητέ ανακαλύπτουν ότι όταν ζητήσουν δουλειά τα προσόντα που έχουν και οι γνώσεις που έμασαν είναι ανεπαρκείς. Και τρίτον, ξέρω και είναι απογοητευτικό για τη χώρα μου ότι τα καλύτερα πανεπιστήμια υποβασμίστηκαν στην αξιολόγηση, στο ranking δηλαδή και έπεσαν στη σειρά του καταλόγου αξιολόγησης. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους ομιλητές να μας πούν τη γνώμη τους. Τι πιστεύουν για αυτή την κατάταξη, για αυτό το κατάλογο κατάταξης και αξιολόγησης, εάν είναι σωστό να γίνεται, αν ξέρουν με ποιο τρόπο γίνεται και αν πιστεύουν ότι θα πρέπει να ε, διοχετεύονται οι πιστώσεις και τα χρήματα στα καλύτερα πανεπιστήμια ανάλογα με την κατάταξή τους. Ε, πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή μας και αυτό το φόρουμ είναι το κατάλληλο για να θέσω αυτή την ερώτηση. Όλοι θέλουμε να είναι μια σωστή κατάταξη των πανεπιστημίων. Σίλβια κυρία πολύ χρήσιμη αυτή η ακρόαση έτσι ώστε να δοθεί μία συνέχεια στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Γιατί θα πρέπει να προβάλλουμε και μία πολυφωνία με βάση αυτή την ανακοίνωση. Μιλάμε για τη διαβίου μάθηση και μιλάμε για το ανθρώπινο δυναμικό, για το ανθρώπινο κεφάλαιο μέσα στα πλαίσια και της διαδικασίας της Μπολόνια, η οποία θα πρέπει να επανειδωθεί υπό αυτό το φως, δηλαδή των ευκαιριών που μπορεί να έχει ο άνθρωπος μέσα στα πλαίσια της κατάρτισης και του εργασιακού περιβάλλοντος. Και όπως είπε και ο υπεύθυνος, του Φιλανδικού Ινστιτούτου, μέσα στα πλαίσια αυτού του τριγώνου των γνώσεων, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος δεσμός μεταξύ εκπαίδευσης, νοτομίας και έρευνας. Και αυτό βοηθάει στην απασχολησιμότητα. Άρα τα πανεπιστήμια με βάση τη διαδικασία της Μπολόνια θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας αξιολόγησης και να δοθεί μια όθηση έτσι ώστε να εγγυηθούμε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα στον άνθρωπο και να μπορούν να μεταφερθούν αυτές οι γνώσεις, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν αδύναμο κρίκο του συστήματος. Συμμετείχα σε μία ακρόαση για τις ε, καινοτόμους υπηρεσίες όπου λένε, ακριβώς ανέφεραν, ότι δυστυχώς ε, δεν μπορεί να γίνει η μετάβαση μεταξύ πανεπιστημιακής έρευνας στην εφαρμοσιμότητα δηλαδή στην έμπρακτη εφαρμογή. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε μια πολιτική στρατηγική έτσι ώστε να αναπτυχθούν αυτοί οι δεσμοί μεταξύ πανεπιστημίων ε, και έρευνας με την απασχολησιμότητα. Επίσης, ως προς την κινητικότητα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτό αυτά τα προσόντα, διότι αυτό που έχει σημασία να δούμε ότι στο έρασμος υπάρχουν οι νέοι φοιτητέ αλλά και οι νέοι επιχειρηματίες. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη δύο προτάσεις, δηλαδή στις παραμέτρους αξιολόγησης των πανεπιστημίων σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκής αξιολόγησης να βλέπουμε την ποσότητα και την ποιότητα κινητικότητας φοιτητών διδασκόντων, μεταφορά της γνώσης και συμμετοχή στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Μιλάμε για διαβίου μάθηση και για διαρκή μάθηση. Δεν ξέρω πώς έχει ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο, διότι θα πρέπει ε, να υπάρχει ε, πρόσβαση σε υψηλό επίπεδο απόκτησης γνώσεων κατά τη διάρκεια και του επαγγελματικού βίου μέσα στα πλαίσια της ε, διαρκούς γνώσης και να προβάλλουμε εταιρικές ε, σχέσεις κατάρτισης στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις. Αναθεματικές ενότητες χρησιμοποιώντας ε, και το, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με βάση ε, ευέλικτα σχήματα γνώσης, δηλαδή να μην επίκεντρο μόνο το πανεπιστήμιο, αλλά να υπάρχει και η διαρκής εκπαίδευση, όχι στρίκτο σένσου, αλλά υπό την ευρία έννοια, δηλαδή σε σχέση με την κατάρτιση των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άκουσα τα όσα είπε ο κύριος Σάλιβαν. Και σκέφτηκα το εξή. Οι περισσότεροι μίλησαν αγγλικά, γαλλικά. Θα ήταν καλό να ακούμε και άλλε γλώσσε. Ουγγρικά, σλοβενικά κτλ. Υπάρχουν βέβαια κάποια γιατί τα αγγλικά μιλούνται παντού στην Ευρώπη. αλλά δεν δίνουμε την κατάλληλη έμφαση ή ανάλογη έμφαση στις μικρές γλώσσες. Το Erasmus είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει στεφθεί με επιτυχία. Έχω συγκινήσει οι οποίοι έχουν ε, συμμετάσχει στο πρόγραμμα Εράσμους στη Γερμανία, στην Αγγλία και γνωρίζω το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στην γλωσσική πολυμορφία. Και όσον αφορά τους Ούγγρους φοιτητέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στο πρόγραμμα αυτό, αλλά να καταφέρουμε να προωθήσουμε μέσω του προγράμματος αυτού και τις α, μικρές γλώσσες. Θα ήταν σημαντικό να μπορούμε να έχουμε προγράμματα όπως το Εράσμους και σε γλώσσες όπως η δικιά μου, τα Ουγγρικά, δηλαδή να προωθούν περισσότερες μικρές γλώσσες. Ich glaube, es ist Νομίζω ότι κάποια παρανόηση έχει γίνει με το Εράσμος, με αυτά που βλέπω εδώ. Η κυρία Σάλιβαν, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους προλαλήσαντες ε, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση ε, που ε, γίνεται βάση και λόγω της ανακοίνωσης της Κομισιόν. Από ό,τι ήξερα, ο στόχος ε, της διαδικασίας της Μπολόνια και όλης της τροβάσμιας εκπαίδευσης είναι να αυξήσει και να ενισχύσει την κινητικότητα, που είναι μια θαυμάσια ιδέα. Όλοι συμφωνούμε, όλοι θα υποφεληθούν από αυτή την αυξημένη κινητικότητα. Όμως υπάρχουν ακόμα σημαντικά προσκόμματα τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Υπάρχει καταρχάς όλο το θέμα των προσόντων και ειδικά του bachelor και η ανάγκη αλλαγής ε, που είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί και ε, η ανάγκη αναγνώριση σε χώρες που δεν το έχουν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάνοντας αυτό το πτυχίο έχεις μια θαυμάσια ε, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά συνδέεται με δυσκολίες Εν συνεχεία υπάρχουν οι γλωσσικές, ε, τα γλωσσικά προβλήματα. Όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια πανευρωπαϊκή ιδέα, σκοντάφτουμε πάντοτε στο γλωσσικό ζήτημα και δεν έχουμε βρει λύση πώς θα το ξεπεράσουμε. Για τους Βρετανούς υπηκόους είναι εύλογο ότι δεν θέλουν να μετακινηθούν εύκολα, δεν θέλουν να αλλάξουν και να πάνε σε άλλη χώρα. Ε, και βεβαίω άλλοι από άλλε χώρες, άλλοι φοιτητέ, ανησυχούν για, για το σε ποια γλώσσα θα γίνει η εκπαίδευση. Και, ε, πρέπει πιστεύω τα γλωσσικά εμπόδια, την προσφορά ε, εκπαίδευση σε ορισμένες γλώσσες, όλα αυτά τα θέματα να τα μελετήσουμε πολύ περισσότερο, διότι πιστεύω ότι η γνώση, η μη γνώση ορισμένων γλωσσών ε, εμποδίζει την κινητικότητα. Το τρίτο πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Πανεπιστήμια στην Ευρώπη έχουν διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης. Το διαπιστώνουμε αυτό όταν μελετήσουμε την χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη. Ε, παραδείγματος χάρη τώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλονται δίδακτρα ε, για, τους, ε, ε, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δεν ξέρω που τι γίνεται ακριβώς σε άλλες χώρες. Δεν λέω ότι όλη η εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν ή να χρηματοδοτείται από το, το δημόσιο, αλλά πρέπει να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν και τι, τα οποία οφείλονται στην επιβολή διδάκτρων ή στο κόστος γενικά. Επίσης, δεν υπάρχει αρκετή επιστημονική κινητικότητα σε επιστημονικούς κλάδους. Πιστεύω ότι και αυτό πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Ε, ένα από τα σημαντικά πράγματα που μπορούμε να επιτύχουμε με την αύξηση της κινητικότητας είναι η βελτίωση της καινοτομίας και της επιστημονικής έρευνας. Αυτό δεν νομίζω να συμβαίνει πουθενά και είναι ένα σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική πτυχή. Επιστημονική κινητικότητα. Σύμφωνο απόλυτα με τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν στην αξιολόγηση. Πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν τρόπο αξιολόγησης ε, και έτσι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την κατάσταση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους ε, τους ε, ομιλητές ε, για τα ενδιαφέροντα σχόλιά τους. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Σε σχέση με τον τελευταίο ομιλητή, μας ενδιαφέρει η επανεισδοχή στο Πανεπιστήμιο των Πρεσβύτερων, να το πούμε, και επειδή υπάρχει η κρίση την οποία διανύουμε, ίσως πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να επανέλθουν στο Πανεπιστήμιο να ε, μπορέσουν να διευρύνουν στη, τις γνώσεις τους. Αλλά τι μπορεί να γίνει σε αυτήν την περίπτωση, πόσο μπορούν να επανενταχθούν, μπορούν να επανενταχθούν με τους νέους, πώς θα είχε αυτή η συμβίωση μεταξύ νεωτέρων και πρεσβυτέρων και τι θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε και οι πρεσβύτεροι να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο Πανεπιστήμιο. Επίσης μιλήσαμε για το ranking των ε, πανεπιστημίων. Είχα διαβάσει νομίζω ότι μεταξύ των 500 πρώτων πανεπιστημίων υπήρχαν μόνο τέσσερα πανεπιστήμια, δηλαδή το Oxford, Cambridge και άλλα δύο αγγλικά πανεπιστήμια. Αυτό ήταν το διεθνές ranking, το οποίο είναι πολύ απογοητευτικό για την Ευρώπη. Δεν ξέρω κατά πόσο το ranking έχει γίνει σωστά ή εμείς ε, δεν τα καταφέρνουμε πράγματι τόσο καλά. Και απαντώντας στον συνάδελφο Ζόλταν για τις ε, γλώσσες. Εγώ μιλώ και ισπανικά και καταλανικά. Πιστεύω όμως, και αυτό το βλέπω και στην πόλη μου, στη Βαρκελόνη, ότι στα πανεπιστήμια μας ε, ε, προσπαθούμε να διδάσκουμε και στα καταλανικά, αλλά πολλοί φοιτητέ από τη Λατινική Αμερική δεν θέλουν να ενταχθούν σε αυτά τα μαθήματα. Γι' αυτό πολύ λιγότεροι μαθαίνουν καταλανικά καθηγητές εννοώ για να διδάξουν στα πανεπιστήμια. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τις μειονοτικές ε, ε, γλώσσες και σε επίπεδο πανεπιστημίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, χρησιμοποιώ όπως ακούτε την συγγενή γλώσσα μου προς τα Ουγγρικά που είναι τα Φιλανδικά. Είναι συγγενής με τα Ουγγρικά. Ε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τα σχόλια, τις ερωτήσεις. Ε, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε η Ευρώπη είναι μια γυραιά ήπειρος και αυτό ε, που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η απασχόληση. Το τρίγωνο αυτό που μας παρουσίασε ο κύριος Μάτιλα είναι η ουσία της υπόθεσης. Και με το τρίγωνο αυτό μπορούμε να βρούμε και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και καινοτόμοι. Βεβαίως χρειαζόμαστε καινοτομία. Έχουμε και ένα λαμπρό παράδειγμα μέσα στην Ευρώπη. Οι παλιές καινοτομίε δεν επαρκούν. Χρειαζόμαστε συνεχώς νέα πράγματα, νέες καινοτομίε. Η Nokia είναι φιλανδική εταιρεία μεταφέρθηκε από τη Γερμανία στη Ρουμανία. Οι εγκαταστάσεις της από τη Γερμανία πήγαν στη Ρουμανία. Πιστεύαμε ότι έτσι θα εξοικονομήσουμε κόστος. Όμως αυτό απέτυχε ε, διότι οι καινοτομίε δεν δούλεψαν στη Ρουμανία. Τώρα κλείνουν και τα εργοστάσια, οι μονάδες στη Ρουμανία. Άρα λοιπόν αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι οι παλιές τεχνολογίες, οι παλιές καινοτομίες δεν επαρκούν. Χρειαζόμαστε συνεχώς καινούργια πράγματα. Η Ευρώπη έχει 27 κράτη-μέλη, διαφορετικές ε, πολιτιστικές πραγματικότητες και διαφορετικά επίπεδα. Είναι πολυεπίπεδη τώρα η Ευρώπη. Εμείς μιλάμε και επισημούμε τη συνεργασία των πανεπιστημίων. Ε, είναι εφικτό αυτό ρεαλιστικά η ισχύ, η δύναμη της ε, ε, Ευρώπης μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητος μας αναγκάζει να, αναρωτηθούμε πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η ενιαία, το ενιαίο επίπεδο, η ενιαία πλατφόρμα ε, και εδώ βλέπουμε συνέχεια ότι τα πανεπιστήμια ενεργούν προστατευτικά, θέλουν να προστατεύσουν την ερευνά τους, τις καινοτομίες τους, ε, τη δουλειά τους, ε, το ακαδημαϊκό τους κύρος ε, και δεν είναι πάρα πολύ πρόθυμα στη συνεργασία αυτή. Ε, πολλά πανεπιστήμια ε, το μόνο που επιδιώκουν είναι να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους. Ε, απεγνωσμένα προσπαθούν να βρουν λεφτά για να μην καταρρεύσουν. Και πολλές φορές αναγκάζονται να συνεργαστούν ας πούμε, με εταιρείε, δεν ξέρω τι, με ερευνητικά προγράμματα για, την, για να βρουν λεφτά. Το θέμα είναι να βρούμε ποια είναι η βέλτιστη πρακτική, πώς μπορούμε να οργανώσουμε αυτή τη συνεργασία στις νέες καινοτομίες. Η πανεπιστημιακή συνεργασία για τις νέες καινοτομίες μπορεί να μας οδηγήσει σε σωτήριες λύσεις. Η Πρόεδρος, ε, δεν ήσασταν και πολύ πιο σύντομα από τους προηγούμενους. Η κυρία Μπενεραμπατού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζούμε σε έναν πολύπλοκο κόσμο με πολλαπλές κρίσεις. Για μένα το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ήταν ένας χώρος όπου θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση είτε είμαστε νέος φοιτητής, είτε είμαστε άνεργος είτε νήλικας. Θα έπρεπε να μπορούμε να μπούμε εύκολα από το Πανεπιστήμιο και να αποφοιτήσουμε εύκολα από το Πανεπιστήμιο. Ο κύριο Φετρή μα μίλησε για τη διαβίου μάθηση και πιστεύω ότι πραγματικά αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο. Και εγώ αυτό ακριβώς έκανα στη ζωή μου. Πολλές φορές σε διάφορα στάδια της ζωής μου εγγράφηκα στο πανεπιστήμιο και αποφύτησα από το πανεπιστήμιο με βάση τις ανάγκες που είχα κατά καιρού. Η κυρία Παλιαδέλη αναφέρθηκε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι ανθρωπιστικέ επιστήμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Είμαστε, ζούμε σε ένα πολύ δύσκολο, πολύπλοκο κόσμο που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Όταν παίρνουμε το πολιτήριό μα και πάμε στο πρώτο έτος του πανεπιστήμιου, ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο δρόμο, κάνουμε μια επιλογή και μετά από πέντε χρόνια συνειδητοποιούμε ότι έχουμε επιλέξει σπουδέ οι οποίε είναι παροχημένε και βλέπουμε ότι στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι οι οποίοι είναι άνεργοι. Νέοι οι οποίοι επέλεξαν κάποιε πανεπιστημιακέ σπουδέ και νέοι οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι από την αρχή των σπουδών του, μέχρι το τέλο των σπουδών του, η επιλογή που είχαν κάνει ήταν παροχημένη είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την παραδοσιακή αυτή προσέγγιση και αντιμετώπιση των σπουδών. Δηλαδή ότι αποφυτώ από το σχολείο, μπαίνω στο πανεπιστήμιο, κάνω ένα πτυχίο και μετά πιάνω δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προσδώσουμε στου νέου αυτού, τι απαραίτητε δεξιότητε, προκειμένου να βρουν μια θέση εργασία. Τα πράγματα όμω είναι πιο πολύπλοκα το θέλουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πανεπιστήμιο όπου θα μπορούν οι άνθρωποι να εγγράφονται και να αποφυτούν ανα πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Και έπειτα το θέμα της αξιολόγηση είδους αξιολόγηση μπορούμε να κάνουμε. Αν η αξιολόγηση ουσιαστικά περιορίζεται σε μία κατάρτιση, η οποία θα βασίζεται μόνο στις ε, επιδόσεις που έχουν τα πανεπιστήμια συγκεκριμένα για τον επαγγελματικό τομέα, τότε πραγματικά δεν προχωρούμε σωστά. Δεν θα πρέπει τα πανεπιστήμια να αξιολογούνται μόνο με βάση τις θέσεις απασχόλησης, επαγγελματικές επιδόσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα πανεπιστήμια να είναι λίκνα γνώσης. Για παράδειγμα, στο Παρίσι Υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές σχολές όπως η Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ή η Σχολή Φιλοσοφίας. Είναι χώροι που μπορεί κανείς ε, να παρακολουθήσει μαθήματα χωρίς να έχει εγγραφεί επίσημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε ακριβώς να αποφεληθούμε τις γνώσεις αυτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επομένως να δούμε ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την κατάταξη του πανεπιστημίων. Λυπάμαι που το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει σε μια παροχημένη προσέγγιση πανεπιστημίων και αναφέρεται μόνο στη διασύνδεση του πανεπιστημίων και του χώρου εργασίας. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλού πτυχιούχου πλέον οι οποίοι είναι άνεργοι. Μόνο και μόνο αυτό θα πρέπει να μα ταράξει λίγο, να μα κάνει να ρωτηθούμε. Κάνουμε σωστά τα πράγματα. Έχουμε σκεφτεί σωστά τα πράγματα. Αν έχουμε τόσου πολλού οι οποίοι είναι σωστά καταρτισμένοι κατά τα άλλα. μήπω θα πρέπει να ξαναδούμε την όλη διαδικασία. μήπω θα πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι χώροι όπου διαμορφώνουμε όχι μόνο μελλοντικού εργαζομένου, αλλά και συντοποιημένου πολίτε. Πιστεύω ακριβώ ότι ε, οι ανθρωπιστικές επιστήμες θα μας επιτρέψουν να έχουμε το πολιτιστικό αυτό υπόβαθρο, το οποίο θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω δύο παρατήρησει. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Ιταλό καθηγητή, ο οποίος είπε ακριβώς αυτό που πιστεύουμε εμείς, ότι με το bachelor εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ε, τα αγγλικά πανεπιστήμια δίνουν το bachelor και όταν ε, ήμουνα στο Göteborg και ρώτησα ε, πώς το κάνετε, τέλος πάντων πώς το εφαρμόζετε, μου είπαν ότι πάντοτε είχαμε έναν υποψήφιο και ένας υποψήφιος ήταν ακριβώς αυτός που είχε ένα bachelor. Δηλαδή είχαν μία υποδομή την οποία δεν είχαμε εμείς και το bachelor στην Μεγάλη Βρετανία μπορεί να έχει επαγγελματική αξία, αλλά στις άλλες χώρες ε, εξαπολιέται ο, ο, ο καημένος, ο κάτοχος του bachelor να βρει δουλειά και δεν μπορεί διότι κανένας δεν τον χρειάζεται, κανένας δεν έχει τη δυνατότητα να τον απασχολήσει. Πρέπει λοιπόν το ακαδημαϊκό, η ακαδημαϊκή ηγεσία να προσπαθήσει να ρυθμίσει αυτό το θέμα του bachelor και της ε, αξιολόγησης του στην ιεραρχία των ε, πτυχίων. Κάτι έχει διορθωθεί, αλλά πολύ λίγο. Μόνο τα πανεπιστήμια μπορούν να το ρυθμίσουν αυτό, ούτε βουλευτές, ούτε πολιτικοί. Λοιπόν, αυτό είναι πήγον. Δεύτερο, η αξιολόγηση, το ranking. Το ranking το οποίο ξέρουμε εμείς είναι το, η αξιολόγηση της αριστείας. Ε, και έχουμε και ένα γλωσσικό πρόβλημα. Αυτή η πολυγλωσσία στην Ευρώπη είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη της αριστείας και της καλύτερης ε, βαθμολογίας εγώ που κατάλαβα την Κομισιόν καλύτερα από την ε, συνάδελφο Μπεναράμπα του, η, η Κομισιόν έχει ένα καλύτερο σύστημα. Θέλει να κατατάξει καταρχάς, να ομοδοποιήσει τα πανεπιστήμια ανάλογα με την ειδίκευσή τους. Ποια πανεπιστήμια κάνουν αυτό καλύτερα ή το άλλο καλύτερα ή τα για να μπορούμε να είμαστε σοβαροί, να εφαρμόσουμε σωστά κριτήρια και να πούμε ότι αυτά τα πανεπιστήμια είναι καλύτερα. Όχι μόνο στην έρευνα, αλλά και στη διδασκαλία. Εάν δεν λάβουμε υπόψη και αν δεν δώσουμε προτεραιότητα στη διδασκαλία, στο ranking θα είμαστε πάντοτε χαμηλά. Επίσης, χαίρομαι ιδιαίτερα που ο τελευταίος ομιλητής για τη διαβίω εκπαίδευση είπε αυτό που λέμε από την αρχή αυτής της θητείας μας. Ότι δηλαδή η διαβίω εκπαίδευση, η διαβίω εκπαίδευση είναι ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τα πάντα. Από τη γέννηση μέχρι το θάνατο του ατόμου. Τώρα θέλουν ε, κάπου στους διαδρόμους και στις πίσω αίθουσες ε, θέλουν να βρουν μια καινούρια προσέγγιση και να καταργήσουν τον όρο lifelong learning, διαβίω εκπαίδευση. Όμως είναι τόσο σημαντική αυτή η έννοια που επιτέλους καταφέραμε να αναγνωριστεί ώστε εάν καταργηθεί και αν τη σβήσουμε θα την πατήσουμε άσκημα. Γι' αυτό σας παρακαλώ ε, μέχρι τις 23 ε, να, να, να, εκφράσετε την άποψή σας, να ακουστεί η φωνή σας ότι αυτό δεν είναι σωστό, είναι μεγάλο σφάλμα. Τόσα χρόνια παλεύαμε για να βρεθεί ο όρος LLL, Lifelong Learning. Τώρα θέλουν να τον εξαφανίσουν, να τον σβήσουν. Κάτι γίνεται, κάτι μαγειρεύεται και δεν ξέρουμε τι. Κάτι ακόμα. Κάποιος είπε ότι το Erasmus Mundus έχει μικρή συμμετοχή. Σας θυμίζω, το Erasmus Mundus ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο θα άνοιγε τις πόρτες τις δικές μας προς όλο τον κόσμο. Τώρα έχουμε επιτύχει και το αντίθετο, ότι όσοι κάνουν διδακτορικό στην Ευρώπη, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να κάνουν το διδακτορικό τους και σε άλλες χώρες, σε τρίτες χώρες. Γιατί τώρα αυτή η μικρή συμμετοχή. Βέβαια, ένας λόγος είναι ότι λίγοι συμμετέχουν επειδή δεν έχουμε ακόμα τόσα πολλά χρόνια. Κάποιος άλλος μίλησε για το πρόγραμμα Bonus, ανατολικό Α, το πρόγραμμα της Βαλτικής θάλασσας. Δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό. Ίσως μπορέσετε να μας φωτίσετε λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω ποιο πρόγραμμα είναι αυτό. Και τώρα παρακαλώ τους ε, εμπειρογνώμονές μας να απαντήσουν. Ό, ό, όσο μπορούν πιο σύντομα, παρακαλώ. κύριος Λούτσατ, <laughs> πρώτος. Uh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Θα αναφερθώ σε τρία σημεία, τα οποία αποτελούν περισσότερο αντικείμενο της αρμοδιότητάς μου. Με συγχωρείτε. Εκτός μικροφώνη, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, απαντά ο μιλητής. Το πρώτο θέμα εφήγει από την ε, πρόεδρο που αφορά τα bachelor. Βεβαίως η κατάσταση στη Γερμανία και στην Ιταλία είναι παράλληλη και αυτό αφορά τους ακαδημαϊκούς μας, διότι αυτό ε, σχετίζεται και με το γεγονός ότι οι καθηγητές της Γερμανίας και της Ιταλίας θεωρούν ότι έκαναν ό,τι καλύτερο και δεν υπάρχει τίποτα που θα όφιλε να αλλάξει. Δεν είναι μόνο πρόβλημα των πανεπιστήμιων. Θα πρέπει να βρούμε και συνοδευτικά θεσμικά και πολιτικά μέτρα σε σχέση με τη χρήση των τίτλων στο δημόσιο τομέα. Είναι ένα θέμα που ήταν αποφασιστικής σημασίας και αυτό το έθεσε και ο κύριος Βίγκλερ στη Βιέννη. Θα πρέπει να διανύσουμε πολύ δρόμο και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ε, επαυξήσουν την ε, χρησιμότητα των bachelor. Θα πρέπει να αλλάξουν δηλαδή. Και θα ήθελα να πω ότι θα σας ε, αποστείλω έγγραφα, αν μου το επιτρέψει η πρόοδος, που δείχνουν ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε τόσο πολύ για τα Bachelor. Μία γερμανική ομάδα από τον κύριο Τάιχνερ ανέλαβε αυτό το έργο και έδειξε ότι και εκεί που δεν υπήρχε υπάρχει αυτή η θέληση των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το bachelor και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχουν ε, δηλαδή προκαταλήψεις ως προς αυτό το θέμα. Δεύτερον, το θέμα των αξιολογήσεων, το ranking. Αυτό θίγει πλιστάκης και θα πρέπει να μας απασχολήσει και εδώ, διότι Σίγουρα, ακόμα και αν ε, επικρίνουμε πάντα, θεωρούμε ότι τα, ε, τα κριτήρια δεν είναι πάντα αντικειμενικά και ενδεχομένως ίσως ε, δεν υπάρχουν πάντα αντικειμενικά δεδομένα. Πολλοί μπορούμε να ασφάλουμε, αλλά μας ενδιαφέρουν τα κριτήρια, οι παράμετροι που λαμβάνουμε υπόψη στα rankings. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία και δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε, διότι πολλές φορές γίνεται για διαφάνεια και όχι για rankings. Ε, αυτό όμως δεν είναι σωστό, γιατί αν τα rankings υπάρχουν αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη, τότε τι κάνουμε. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι παράμετροι που χρηματοδοτεί και η Κομισιόν και θα πρέπει να δούμε τι, ε, ποια είναι η αποστολή των πανεπιστημίων έτσι ώστε να υπάρχει μία ομογενειοποίηση των κλάστερς πανεπιστημίων. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο να βάλουμε υπόψη την έρευνα ή και άλλες αξίες. Δηλαδή, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία εκπαίδευσης. Ας δούμε τα αποτελέσματα των πτυχιούχων, όχι τον αριθμό τους, τα αποτελέσματά τους. Τα αποτελέσματα, έτσι θα κρίνουμε τα πανεπιστήμια. Δεν είναι εύκολο ε, και δεν είναι εύκολα μετρήσιμα τα αποτελέσματα των πτυχιούχων ελέγχθη ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ληφθούν υπόψη μόνο τα μετρήσιμα στοιχεία. Ε, όμως θα πρέπει να δούμε την ουσία και όχι την μετρησιμότητα όλων των στοιχείων. Να δούμε το ρόλο των πανεπιστημίων όχι μόνο για τα 3L, αλλά και τη σχέση των πανεπιστημίων με την κοινωνία τη σχέση με τους πολίτες. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση. Ε, Mr. Ο κύριος Σάλιβαν, σας ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση αυτή είναι πραγματικά η πλέον κατάλληλη και ιδιαίτερα σημαντική. Πρέπει να σας πω ότι διανύουμε μία από τις χειρότερες οικονομικές βιομηχανικές κρίσεις της Ευρώπης που έχει προκαλέσει πολλά κοινωνικά και πολιτιστικά προβλήματα. Ωστόσο εξακολουθούμε και έχουμε τον πιο καταρτισμένο πολιτισμό, πληθυσμό που είχαμε ποτέ στην ιστορία της Ευρώπης. Και ξέρετε ότι ακόμα και πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν προκαλέσει τα προβλήματα της κρίσης αυτής είναι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας. Επομένω, καλούμαστε αυτή τη στιγμή να δούμε ακριβώς τον ρόλο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όσον αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών αυτών προκλήσεων. Να αναφερθώ καταρχάς στο ζήτημα του ranking της α, ταξινόμησης. Νομίζω ότι αποτελεί αιμονή για πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν 4.000 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εράσμους. Οποιοδήποτε σύστημα και ranking να χρησιμοποιήσει κανείς, κάποιο τελικά θα βρίσκεται πάντα στου πρώτου 100. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν είναι καλά, ότι δεν καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους, ότι δεν επιφέρουν μια προστιθέμενη αξία για όσου εργάζονται και φοιτητούν στα, σπουδάζουν στα ιδρύματα αυτά. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, τα ranking έχουν ως κύριο στόχο το output, το αποτέλεσμα. Έχουμε ένα διτό σύστημα στην Ιρλανδία, όπου έχουμε τα τεχνολογικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια. Τα τεχνολογικά ιδρύματα ξεκίνησαν το 1960, εκείνη τη δεκαετία, και ουσιαστικά ανταποκρίθηκαν σε μια νέα προσέγγιση της οικονομίας στην Ιρλανδία. Από μια προστατευόμενη κλειστή οικονομία περάσαμε σε ένα σύστημα πιο ευέλικτη, ανοιχτής οικονομία Τα τεχνικά λοιπόν αυτά ιδρύματα έχουν φοιτητέ οι οποίοι ενδεχομένω έχουν ένα χαμηλότερο επίπεδο όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χαμηλότερου βαθμού και παρόλα αυτά καταλήγουν με πτυχιούχου οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι, οι οποίοι βρίσκουν πολύ καλέ θέσει εργασία και συμβάλλουν πάρα πολύ στην εργασία του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για αυτόν τον λόγο η Ιρλανδία είναι ιδιαίτερα ελκυστική και όχι μόνο επειδή έχει χαμηλό εταιρικό φόρο. Ουσιαστικά δίνουμε μέσω του συστήματός μας ευκαιρίες στους ανθρώπους, οι οποίοι διαφορετικά θα πρέπει να είχαν μεταναστεύσει, δεν θα είχαν τις ίδιες επαγγελματικέ ευκαιρίες με αυτές τις οποίες τους προσφέρουμε. Αν ρωτήσετε έναν εργαζόμενο πλέον απόφυτο από τα τεχνικά αυτά ιδρύματα σχετικά με τα rankings θα σας πούνε ότι σίγουρα εγώ δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση που πήγα σε ένα τεχνολογικό ίδρυμα, μάλλον ότι μπορεί να με βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στα ranking. Ετέθηκε ένα ερώτημα που είχε να κάνει με την ευθυγράμμιση των πανεπιστημίων, των ε, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις ανάγκες του, της αγοράς εργασίας. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει ακριβώς κανείς ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, ποιες είναι οι ανάγκες του βιομηχανικού κλάδου χρειάζονται βασικά τέσσερα πράγματα. καταρχά, ευελιξία, δημιουργικότητα, τη δυνατότητα εργασία στα πλαίσια μια ομάδα και δυνατότητα επικοινωνία. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που ζητάει η αγορά εργασία. Και γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια τη παρουσίαση μου, μου, αναφέρθηκα στην κινητικότητα. Πιστεύω ότι η κινητικότητα μπορεί να συμβάλλει στο να κερδίσει κανεί αυτά τα χαρακτηριστικά. Και δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για δεξιότητε. Σαφώ μπορούμε να μάθουμε σε κάποιον πώ να χρησιμοποιεί ένα υπολογιστή, αλλά πώ μπορεί να μάθει κανεί σε κάποιον να να επινοεί έναν υπολογιστή, να δημιουργεί έναν υπολογιστή. Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να συνδέσουμε καλύτερα τα πανεπιστήμια με το χώρο εργασίας. Χρειαζόμαστε αυτές τις συνεχείς διαρκείς δεξιότητες, οι οποίες προέρχονται περισσότερο τελικά από τη διαφύου μάθηση. Και αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι να έχουμε εκπαιδευόμενους οι οποίοι αργότερα στη ζωή τους θα θελήσουν να επιστρέψουν στα πανεπιστήμια ή σε κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους. Ουσιαστικά αυτούς τους φοιτητές θα πρέπει να προωθήσουμε και αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να προωθήσουμε. Θα μπορούσατε ουσιαστικά να αναφερθείτε σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη τέτοια προγράμματα κατάρτισης. Είναι ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές πολλές φορές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν κάποια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Νομίζω ότι ακριβώς αυτές οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να τις βοηθήσουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μάτιλα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, θα χρησιμοποιήσω και εγώ μία μικρή γλώσσα συγγενής προς τα Ουγγρικά. Η κυρία Πρόεδρος έθεσε ένα ερώτημα γιατί μόνο μερικά πανεπιστήμια, ορισμένα πανεπιστήμια είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα του Erasmus Mundus. Αυτά τα διδακτορικά προγράμματα στις διάφορες χώρες και πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και είναι δύσκολο να γίνει η διασύνδεση ε, μεταξύ των πανεπιστημίων για αυτά τα προγράμματα. Το βήμα αυτό είναι βήμα μεγάλης αλλαγής στα πανεπιστήμια και γι' αυτό ακριβώς λίγα πανεπιστήμια συμμετέχουν. Λίγα είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να εκπονήσουν ένα κοινό διδακτορικό πρόγραμμα του που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Εράσμους Μούντους. Δεύτερο ερώτημα. τα υποστημονικά προγράμματα, το, το πρόγραμμα της ε, Βαλτικής θάλασσας ε, είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο άρθρο 185 της συνθήκης. Είναι ένα κοινό πρόγραμμα που το διαχειρίζεται μία, ένας ανεξάρτητος φορέας. Συμμετέχει και η Γερμανία, είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων των χωρών της ε, Βόρειας Θάλασσας, ε, της Βαλτικής ε, κυρίως, στη λήψη των αποφάσεων. Υποστηρίζει αλλά και εκπαιδεύει η σύνοντα στελέχη των χωρών αυτών για τη λήψη αποφάσεων. Θα μπορούσα να σας στείλω πληροφορίες, να σας διαβιβάσω πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα, εφόσον δεν το γνωρίζετε, πληροφορίες και στοιχεία. Και άλλο ένα σχόλιο. Ο κύριος Τάκουλα ρώτησε γιατί γιατί δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε την ανάγκη μιας ε, ε, ε, ευθυγράμμισης, μιας ανόδου το, της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ευρώπης σε ανώτερο επίπεδο, σε, μεγαλύτερο, σε υψηλότερο επίπεδο. Κοιτάξτε, μεταξύ των πανεπιστημίων υπάρχουν ε, δίκτυα βέλτιστης πρακτικής, ε, υπάρχει το LEDU, ε, ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τα ερευνητικά προγράμματα των καλύτερων πανεπιστημίων. Είναι ένα κλειστό δίκτυο αυτό, ένα κλειστό δίκτυο των καλύτερων πανεπιστημίων και έτσι και καλό, γιατί έτσι επιτυχάνονται οι βέλτιστες πρακτικές. Υπάρχει και ένα άλλο δίκτυο συνεργασίας, η Κοϊμπρά, που ονομάστηκε έτσι βάσει της πορτογαλικής πόλης Κοίμπρα. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν παλαιότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, παλαιότερα δηλαδή από την χρονολογία ίδρυσης. Ίσως το δίκτυο αυτό Κοίμπρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Όμως χρειαζόμαστε και άλλα δίκτυα συνεργασίας ε, Πολλά μπορούμε να κάνουμε ακόμη για τη συνεργασία σε υψηλό επίπεδο. Και ο κύριος ο πρόσωπος της Καταλωνίας ρώτησε γιατί τα Αμερικά πανεπιστήμια είναι τόσο καλύτερα από ορισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Όσον αφορά αυτό το, την αξιολόγηση, αυτό το ranking, κοιτάξτε, για να το πούμε απλά, πρώτη για λεφτά. Είναι τα λεφτά, οι πόροι, έτσι ο προϋπολογισμός πολλών Αμερικανικών πανεπιστημίων είναι μεγαλύτερο σε ένα πανεπιστήμιο από τη χρηματοδότηση όλων των φιλανδικών πανεπιστημίων. Ένα Αμερικανικό πανεπιστήμιο έχει περισσότερα λεφτά από όλα τα φιλανδικά. Δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να έχουμε τόσα κονδύλια. Όμως, ορισμένα τμήματα, ορισμένα επιστημονικά τμήματα των πανεπιστημίων στην Ευρώπη έχουν υψίστη αναγνώριση στον κόσμο και πιστεύω ότι ορισμένες μικρές, μικρότερες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά τα δίκτυα αριστείας με τους καλύτερους επιστήμονές τους παρόλο που δεν έχουν τις δυνατότητες των Αμερικανικών. Όσον αφορά τώρα τις γλώσσες, το γλωσσικό πρόβλημα μέσα στα πλαίσια του Εράσμους, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το εξής. Ε, να προσφέρουμε εκπαίδευση στα αγγλικά Έχουμε και φιλανδικά και σουηδικά. Είναι οι δύο επίσημες γλώσσες της Φιλανδίας. Φιλανδικά και σουηδικά. Ε, είναι εύκολο να εκπονήσουμε προγράμματα στα σουηδικά. Τώρα αρχίζουμε και ένα ρώσικο. Ένα πρόγραμμα στη ρώσικη γλώσσα. Οπότε όσοι έρθουν ε, φοιτητές ε, θα, θα μελετήσουν και, τον, ε, και το φιλανδικό πολιτισμό, ας πούμε, και τη φιλανδική γλώσσα. Και τέλος, οι τεχνολογικές καινοτομίες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, αυτός ο κλάδος των καινοτομιών για την ανταγωνιστικότητα. Βεβαίως χρειαζόμαστε και ε, καινοτομίες ε, στον κλάδο ας πούμε τον ε, οικονομικό, βιομηχανικό αλλά και στην κοινωνικές καινοτομίες, στην εκπαίδευση, στην υγεία. Εκεί χρειαζόμαστε, πιστεύω, περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν λόγω της οικονομικής κρίσης και ανατομικές προσεγγίσεις. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ ο κύριος Φετρή, ο καθηγητής κύριος Φετρή. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε τέσσερα σημεία, σε τέσσερις ερωτήσεις. Πρώτον, η διαδικασία της Μπολόνια, τουλάχιστον στην αρχική της φάση, είχε επικεντρωθεί περισσότερο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην οργάνωση του συστήματος. Και αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα κατά την άποψή μου. Η όλη διαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα για να λάβουμε υπόψη μα και άλλε διαστάσει. Πρέπει να αντιστρέψουμε τη διαδικασία πλέον και να δώσουμε περισσότερο χώρο και προσοχή στο άτομο έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, αλλά πιστεύω ότι πλέον θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη θέση που κατέχει ο άνθρωπος στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πώς θα καταφέρουμε να εντάξουμε τελικά, να προσαρμόσουμε την Πολόνια στην ε, συνεχιζόμενη σταδιοδρομία ενός ατόμου, στη μετεξέλιξη ενός ανθρώπου. Δεν θα αναφερθώ στα ranking και στις κατατάξεις, αλλά περισσότερο στα κριτήρια αξιολόγησης των ε, διεθνών υπηρεσιών που υπάρχουν. Αν θέλουμε να σημειώνουμε πρόοδο και αν θέλουμε να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτή την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε κατά νου τη διαβίου μάθηση, πρέπει να αλλάξουμε τα κριτήρια αξιολόγησης σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή τα κριτήρια που χρησιμοποιούν διάφορες διεθνείς υπηρεσίες, αλλά και ευρωπαϊκές. γενικά, για παράδειγμα, θα πρέπει να αναθεωρήσει λίγο τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί. Σήμερα πάντως τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται επικεντρώνται πολύ περισσότερο στα ιδρύματα αυτά καθ' αυτά, στην οργάνωση των ανώτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όχι τόσο πολύ στα διδάγματα, στα αποτελέσματα. Τρίτον, συνειδητοποιούμε ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα όσον αφορά την κινητικότητα και την συμβατότητα ανάμεσα στα διαφορετικά διπλώματα, τους τίτλους και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε πλέον μια κοινή γλώσσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια κοινή γλώσσα που είναι ακριβώς αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας μάθησης και αποκόμισης διδαγμάτων. Στη Γαλλία, βλέποντα το όλο και εκτιμένο που έχουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα με την αναγνώριση πτυχίων από τη μία ή την άλλη χώρα. Βλέπω ουσιαστικά υπάρχουν συγκεκριμένα διδάγματα, μονάδες ακαδημαϊκές, οι οποίες έχουν επιτευχθεί με επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο. Αυτό με ενδιαφέρει και αυτό βλέπω. Πιστεύω λοιπόν ότι στα πλαίσια των πανεπιστημίων και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει ακριβώς, ακριβώς αυτό να πετύχουμε, μια καλύτερη ανάγνωση των διδαγμάτων που προέρχονται από τα πανεπιστήμια ποιε είναι οι εγγυήσει που δίνουν τα πανεπιστήμια προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι τελικά μία γνώση έχει όντω κατακτηθεί. Λαμβάνοντα υπόψη πάντα βέβαια τον τοπικό χαρακτήρα ενό πανεπιστημίου. Τέταρτον, να απαντήσω πιο άμεσα σε ερωτήσεις που ετέθησαν, τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη όσον αφορά την διαβίου μάθηση και τη διαβίου κατάρτιση, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να παραμείνει ένας ανοιχτός χώρος. Σήμερα δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα κοινό μοντέλο. Πειραματιστήκαμε ένα πρώτο διάστημα με ένα μοντέλο που είχε να κάνει με την διαβίω επαγγελματική κατάρτιση που επιμέρους κάποια πανεπιστήμια εφάρμοσαν. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε πολλαπλές και διαφορετικές απαντήσεις, γιατί και οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και οι ανάγκες είναι πολλές και διαφορετικές. ενδεχομένως να φτάσουμε και στο σημείο να υποδεχθούμε σε ένα επιστημονικό εργαστήριο ένα άτομο για μία εβδομάδα, επειδή το άτομο αυτό πρέπει να καταρτιστεί μία εβδομάδα σε μια συγκεκριμένη βιομηχανική ερευνητική διαδικασία. Κάποια άλλη στιγμή θα πρέπει να προσφέρουμε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης τεχνικών γνώσεων, Άλλοτε θα πρέπει να προσφέρουμε προγράμματα που θα έχουν να κάνουν με αναβάθμιση συγκεκριμένων πτυχίων. Α πάρουμε την κινητή τηλεφωνία, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν στον τομέα των σταθερών τηλεφώνων και έπρεπε κάποια στιγμή να καταπιστούν στα ζητήματα τη κινητή τηλεφωνία. Η ε, απάντηση λοιπόν που θα πρέπει να δώσουμε είναι μία απάντηση κατάλληλη, η οποία να μην είναι ουσιαστικά μόνο ένα σύντομο πρόγραμμα μερικών ωρών, αλλά να μπορούμε ουσιαστικά στα πλαίσια της διαβίου μάθησης να καλύψουμε πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Πιστεύω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αναμίξουμε ανθρώπους από πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα άνθρωποι που είχαν την εμπειρία αυτή να έρθουν σε επαφή με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα, ουσιαστικά το έχουν μετανιώσει πολλέ, ποτέ. Υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία υποδέχονται νέους φοιτητές ή ενήλικες ανθρώπους οι οποίοι διεργάζονται και οι οποίοι θέλουν να ξεσκονίσουν κάπως τις γνώσεις τους και έχουμε και πανεπιστήμια που αναπτύσσουν ένα πολύ πιο έντονο και επικοδημητικό διάλογο με αυτούς τους φοιτητές που προέρχονται από διαφορετικές ηλικίε και διαφορετικά περιβάλλοντα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε και το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι θετικό. Ζητάτε όμως πολλά από τους καθηγητές, λέει η Πρόεδρος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην Πολωνία. Να μας μιλήσετε έντονα, αλλά όχι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σας παρακαλώ. Θα μιλήσω πολωνικά, επομένως σας παρακαλώ πολύ τα ακουστικά σας. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Θέλω εξ αρχής να πω ότι εκπροσωπώ το Υπουργείο Σχολικής Εκπαίδευσης, αλλά είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Ούνι που μου δίνει και μια άλλη προοπτική. Η διαδικασία της Μπολόνια και οι αλλαγές στην τριτοβάθμια ευρωπαϊκή εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια καλή ιδέα είναι μία θα έλεγα καθυστερημένη αντίδραση ε, σε διαδικασίες οι οποίες σημειώθηκαν εκτός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το πρώτο γεγονός που επισημάναμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καλά εκπαιδευμένες, ε, για καλά εκπαιδευμένους ε, και φοιτητέ. Ε. Ίσως όχι πάντοτε στο διδακτορικό επίπεδο ή στο επίπεδο του μάστερς, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζεται καλή τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλής ποιότητος. Και πρέπει να διευρυνθεί η στο επιπεδο του μάστερ, αλλα εν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως το είπε και ο Ιρλανδός καλεσμένος. 70% ε, των νέων ε, στην Πολωνία σπουδάζουν τα τελευταία χρόνια πενταπλασιάστηκε ο αριθμό των φοιτητών στην Πολωνία και δεν είναι η μόνη χώρα που έχει αυξήσει τον αριθμό των φοιτητών της τόσο πολύ. Ε, υπάρχει όμως και μια σημαντική θεμελιώδης αλλαγή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εάν θέλουμε τουλάχιστον οι μισοί, ε, μισή νέοι να, να, ε, να, τυχάνουν πανεπιστημιακής μόρφωσης πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στα πανεπιστήμια από την εποχή που το 10% του πληθυσμού σπούδαζε στην βάσμια εκπαίδευση. Η διαδικασία της Μπολόνιας προσπάθησε να βρει ορισμένες απαντήσεις ε, σε αυτά τα προβλήματα. Καταρχάς, ε, καθιέρωσε μία μεταβατική φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν άτομα τα οποία δεν επιδιώκουν ε, το, το μεγαλύτερο πτυχίο να λάβουν μία πανεπιστημιακή μόρφωση μία μεταβατική φάση λοιπόν ε, πρόσβαση στα πανεπιστήμια χωρίς αναγκαστικά απόκτηση του μάστερση του διδακτορικού. Δεύτερον, το θέμα της, ε, του περιεχομένου σπουδών είναι γεγονός ότι όσοι σπουδάζουν τα ίδια χρόνια σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν έχουν όλοι τις ίδιες γνώσεις, έτσι δεν είναι, ούτε τα ίδια μαθήματα, ούτε τα ίδια προσόντα. Από τη μία πλευρά βεβαίως έχουμε αυξήσει την αξιοπιστία των πτυχίων, από την άλλη πλευρά πρέπει να διαμορφώσουμε το περιεχόμενο των σπουδών έτσι ώστε να ταιριάζει στις απαιτήσεις του σπουδάζοντος, του σπουδαστή. Ε, ο σπουδαστής πρέπει να λαμβάνει την εκπαίδευση την οποία θέλει, αλλά ταυτόχρονα και το πτυχίο του να είναι αναγνωρίσιμο και να έχει ουσία. Γιατί? Για να μπορέσουμε να ανταποξέλθουμε στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ε, ε, Φοιτητέ ε, στην Ευρώπη ταξιδεύουν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και ψάχνουν για δουλειά. Είναι μια διασυνοριακή αναζήτηση αυτή και πολλοί από αυτούς βρίσκουν δουλειά στην Γερμανία και σε άλλες χώρες. Τώρα, η αναγνώριση των πτυχίων έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο των σπουδών και με τα προσόντα του φοιτητή. Άρα πρέπει να ε, ξεκαθαρίσουμε τι, θα, ζητούμε από τους φοιτητές και τι ε, περιεχόμενο θα έχει το πτυχίο τους. Αυτό είναι λίγο μια καινούργια προσέγγιση γιατί παλαιότερα τα πανεπιστήμια ήταν κακομαθημένα διότι παίρνανε μόνο τους καλύτερους μαθητές, τους top μαθητές και ήταν ευχαριστημένοι και οι μαθητές και οι καθηγητές με αυτά τα οποία προσφερόντουσαν. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ε, δεν θα πρέπει να μπαίνει μόνο μία ελίτ, αλλά πρέπει να, αυξη... να διευρύνουμε την πρόσβαση ε, και να τονίσουμε και περισσότερο τις ανθρωπιστικές σπουδές. Ε, φιλόσοφοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και, οι και αυτοί δικαιούνται, οι απόφτοι δηλαδή δικαιούνται εργασίας, έτσι δεν είναι πρέπει το ευρωπαϊκό ε, πανεπιστημιακό μοντέλο ε, να ξαναδώσει μεγάλη σημασία ξανά στις ανθρωπιστικές σπουδές. Ε, επίσης, η αναγνώριση των πτυχίων. Έχουμε επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα σωστά, αλλά δεν είμαστε ακόμα, δεν έχουμε φτάσει σε μια τελική λύση. Πρέπει να προσέξουμε το περιεχόμενο των σπουδών, ε, το Πανεπιστήμιο πρέπει να δηλώνει ξεκάθαρα τι επιδιώκει, ποια είναι τα επιτεύγματα και έτσι θα μπορέσουμε να ανεβούμε ποιοτικά. Τώρα, η διασύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας. Δεν συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση ότι με, την ιδέα ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ε, ε, δεν συγκρίνονται με τα αμερικανικά. Δεν νομίζω, διότι οι ρίζες των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων είναι πολύ βασίτερες από τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Μην ξεχνάτε τις ε, ιδέες ε, του Αλεξάνδρ Φον Χούμπολτ, ο οποίος ε, ήθελε να συνδυάσει τους, τη διδασκαλία με την επιστήμη. Αυτά είναι τα θεμέλια των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Διδασκαλία και επιστήμη, διδάσκοντες και επιστήμονες, χέρι με χέρι, να προχωρούν ακαδημαϊκά και έτσι καταφέρουμε να ιδρύσουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν να, ναι, ναι, είναι, είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουν τα, τα πανεπιστήμια τεχνικά ιδρύματα τα οποία προσφέρουν τεχνική εκπαίδευση με πολύ καλό περιεχόμενο, με, με, με πολύ ε, καλά προγράμματα. Αυτό είναι και μια άλλη διχοτόμηση. Δεν, μπορεί να λειτουργούν τελείως ξεχωριστά τα τεχνικά, ας πούμε, οι τεχνολογικά ιδρύματα από τα, τριτο, από την, από τα πανεπιστήμια. Εδώ ζητούμε συνεργασία και συνέργεια, όχι διαχωρισμό. είναι δύσκολο είναι δύσκολο να κρίνουμε ποια πανεπιστήμια προσφέρουν την καλύτερη διδασκαλία, τρόπο διδασκαλίας. Εντάξει, ε, μπορούμε πολύ εύκολα να πούμε ότι οι νομπελίστες της χημίας, της φυσικής και της αστροφυσικής, ας πούμε, προήλθαν από αυτά και αυτά τα πανεπιστήμια. Όμως, αυτό είναι εύκολο να κατατάξουμε τα πανεπιστήμια βάση. Ε, της του επιστημονικού κλάδου και των ε, επιστημονικών πτυχίων που δίνουν. Αλλά τι γίνεται με τη διδασκαλία. Πώς μπορούμε να κρίνουμε το ανθρωπιστικό, τον ανθρώπινο παράγοντα στα πανεπιστήμια. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Βλέποντας, ε, ακούγοντας την ομιλία σας, βλέπω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό σύνδεσμο ε, στην Πολωνία και συμφωνώ απόλυτα με την ανθρωπιστική ε, αξία που δώσατε στους διδάσκοντες και στους ανθρώπους δηλαδή που, που εκτελούν αυτό το ρόλο. Η Κομισιόν, ο κύριος Τάισον. Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά και θα χρησιμοποιήσω τη δικαιολογία ότι είναι η μητρική μου. Πρόκειται για μία ακρόαση για τη διαδικασία της Μπολόνια και πού βρισκόμαστε στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Επίσης, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι η Κομισιόν εξέδωσε τη δική της ανακοίνωση για τον εξυγχρονισμό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δύο εβδομάδες πριν και υπάρχει επικάλυψη γιατί προσπαθούμε στην Κομισιόν να συγχρονίσουμε τις δύο αυτές οδούς, δηλαδή να τις θέσουμε ώστε να κινούνται παράλληλα. Ως προς το ρόλο των ΑΕΗ, θα Ήθελα να πω και να επαναλάβω ίσως ότι ο πρωταρχικός στόχος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η δημιουργία και η διαβίβαση γνώσεων. Και στην Ευρώπη κατέχουμε ε, δεσπόζουσα θέση, προσπαθούμε να το καταφέρουμε αυτό. Και αυτό μέσα στα πλαίσια δημοκρατικών διαδικασιών. Εμένουμε πολύ σε αυτό παρά το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν τα καταφέρουν καλά στα διάφορα rankings. Ε, δηλαδή, ε, μόνο τα 28 ε, γύρω στα 28 από τα 140 βρίσκονται σε καλό επίπεδο αξιολόγησης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανησυχούμε, και σας συστήνω να ρίξετε μια ματιά στην αξιολόγηση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι. Συμφωνώ όμως με τον καθηγητή Μάτιλα ότι υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αξιολόγησης των πανεπιστημίων και του επίπεδου επενδύσεων από πλευράς ε, ως προς την έρευνα. Δηλαδή βρισκόμαστε κάτω από το 3% του ΑΕΠ στο οποίο έχουν προσυπογράψει τα κράτη-μέλη για τη χρηματοδότηση στην έρευνα. Ο καθηγητής Μάτιλα επίσης έκανε μία σύγκριση μεταξύ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ και των Φιλανδικών Πανεπιστημίων. Αλλά η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Το Χάρβαρτ είναι το πιο πλούσιο πανεπιστήμιο στον κόσμο και έχει ένα ιδιωτικό ταμείο που χρηματοδοτεί όλες του τις δραστηριότητες. Το μέγεθος είναι σαν ολόκληρη την κερδοφορία όλων των ΑΕΗ στην Ευρώπη. Δηλαδή η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας όταν το χάσμα είναι τόσο μεγάλο. Και αφορά ιδιαίτερα το, ε, τον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι δημόσιες επενδύσεις είναι στο ίδιο επίπεδο με τον ΙΠΑ. Δηλαδή βρισκόμαστε στα ίδια περίπου επίπεδα. Για να επανέλθω στην Πολόνια, ξεχνάμε πολλές φορές ότι η Πολόνια τα πρώτα 10-11 χρόνια προέβαλε μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Τα δύο τρίτα των 47 κρατών που καλύπτονται από την Πολόνια ήδη έχουν οργανώσει το 90% των προγραμμάτων τους έτσι ώστε να συνάδουμε αυτή τη διαδικασία bachelor, master και διδακτορικό. Υπάρχουν εξαιρέσεις και εκεί που υπάρχουν αφορούν τα μαθήματα ε, επαγγελμάτων τα οποία βρίσκονται υπό έλεγχο, ελεγχόμενων επαγγελμάτων όπως παραδείγματο χάρη των γιατρών, των ε, νομικών σπουδών και των κτηνιάτρων και ούτω καθεξής. Όμως υπάρχουν χώρες που βασίζονται σε credit 180, άλλες σε 240 και υπάρχει αυτό το διτό σύστημα. Ως προς τον πρώτο κύκλο που οδηγεί στο δεύτερο, το 75% των bachelor ε, δίνουν πρόσβαση σε master, Υπάρχει ένα 25% που αποτελεί πρόβλημα και υπάρχει ε, διαφορά μεταξύ των επαγγελματικών και καθαρά ακαδημαϊκών σπουδών. Ως προς την κινητικότητα έγιναν πολλές επικρίσεις για το σύστημα ECTS, δηλαδή των μεταφορών των credits. Όμως το ECTS χρησιμοποιείται στα 75 5% των μαθημάτων στις 45 από τις 47 χώρες. Άρα μόνο σε δύο χώρες είναι κάτω από 75% αλλά πάνω από 50%. Άρα έχει επιτελεστεί μεγάλη ε, πρόοδος. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Αναφέρθηκα στη δημιουργία των γνώσεων που είναι και ο ρόλος κλειδί των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά ως προς την απασχολησιμότητα, την ανάπτυξη, καινοτομία, ε, ανταγωνιστικότητα και ανάκτηση δυνάμεων από την κρίση, ε, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τους φοιτητές. Αυτό το γνωρίζουμε και γνωρίζουμε ότι με την ανώτατη εκπαίδευση κανείς μπορεί να παραμείνει άνεργος, αλλά διατρέχει λιγότερο κίνδυνο σε σχέση με τη δευτεροβάθμια, σε σχέση με αυτούς που έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως προς την ανταγωνιστικότητα, για να δείτε που είναι η Ευρώπη στον κόσμο, το 2009, αν δείτε το συνολικό αριθμό νέων ε, ε, νέων εισόδων, μάλλον ε, πρόσβαση στην ανώτατη εκπαιδευτικό, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το 1 τρίτον ήταν από την Κίνα. Βλέπετε λοιπόν ότι και η Κίνα, Ρωσία και η Ινδονησία βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στο 3,1% μόνο του προπτυχιακού κύκλου. Θα πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά εισόδου και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη, μεγαλύτερες δυνατότητες εισόδου και άλλοι ε, φοιτητές από την Ευρώπη, το οποίο σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και αυτές οι νέες ομάδες θα πρέπει να εισέλθουν και στο πανεπιστήμιο και στις τεχνικές σχολές, αλλά θα πρέπει να ε, σταματήσουμε την εγκατάλειψη των σπουδών, διότι αρκετοί μπαίνουν αλλά λιγότεροι βγαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μηχανισμούς έτσι ώστε οι φοιτητές που είναι σε μειονεκτούσα θέση να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο. Επίσης η ποιότητα των μαθημάτων έχει σημασία για να μην υπάρχει εγκατάλειψη σπουδών και θα πρέπει να δούμε και νέες ομάδες ε, με τρόπο ώστε να υπάρχει συνδεσιμότητα με τη διαβίου μάθηση. Και έχει μεγάλη σημασία οι ενήλικες να επανέλθουν, οι πρεσβύτεροι ενήλικες. Αν δείτε τις βόρειες χώρες, που βασίζονται στη διαβίου μάθηση βλέπουμε ότι οι δεξιότητες είναι σε καλά επίπεδα σε όλα τα ηλικιακά φάσματα σε σχέση με άλλους, άλλες χώρες της Ευρώπης. Επίσης χρειάζεται καλύτερη συνεργασία με τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να γνωρίζουν οι διδάσκοντες τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Και αυτό δεν σημαίνει ειδικά μαθήματα, αλλά την κριτική σκέψη, την ομαδική εργασία που τους επιτρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία εκμάθησης μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης. Και για να γίνει αυτό πρέπει να ε, προωθήσουμε την αριστεία και στην διδασκαλία και στην έρευνα. Υπάρχουν ε, πριν για την έρευνα, αλλά όχι για, για το διδακτικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν δηλαδή αντισταθμίσεις για τους διδάσκοντες γιατί και για τη σταδιοδρομή αυτό που μετράει είναι η αρθρογραφία, οι εκδόσεις, οι, ε, οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει, αλλά θα πρέπει να γίνει και σε σχέση με το αντικείμενο διδασκαλίας και την πρόθεση συνέργειας με τις επιχειρήσεις. Επίσης, ως προς την περιφερειακή ανάπτυξη θα πρέπει να έχουμε καλύτερες σχέσεις με τις επιχειρήσεις για, τα, για να ενισχύσουμε την αλυσίδα καινοτομίας, τη δημιουργικότητα και να ορίσουμε καλύτερα τις spin-off εταιρείες έτσι ώστε να υπάρχει ένα επίπεδο καινοτομίας, ένα πυρήνας καινοτομίας. Και επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε με θέματα διακυβέρνησης έτσι ώστε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μπορέσουν να δώσουν τα άριστα, αριστότερα δυνατά αποτελέσματα και η χρηματοδότηση να είναι στοχοθετημένη με βάση τις ανάγκες των μεμονωμένων ιδρυμάτων. Ο κύριος Σάλιβαν θα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να υποστηρίξουμε το Dublin Institute of Technology σε σχέση με τα άλλα ιδρύματα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές τους αποστολές. Τέλος, Πρόεδρε, η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των πολιετών χρηματοδοτήσεων πρότεινε να προβούμε σε μία αύξηση της τάξης του 70% και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου. Μάλλον ο μιλτής θα εννοούσε 17%. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στο ε, θέμα της απασχολησιμότητας, κινητικότητας και ούτω καθεξής. και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αυξήσουμε την ποιότητα της κινητικότητας που υποστηρίζει και το πρόγραμμα Εράσμους και το εράσμους Μούντους. Για το Εράσμος Μούντους και γιατί τόσο λίγα πανεπιστήμια συμμετείχαν, ο καθηγητής Μάτιλα έδωσε μία απάντηση. Ο άλλος λόγος είναι τα χρήματα. Υπάρχουν 20 υποψήφοι για κάθε μάθημα του προγράμματος Εράσμος Μούντους Επίσης προβάλλουμε τις συνέργειες γνώσεων, knowledge alliances, με βάση τα διδακτορικά και σας ευχαριστούμε και για τη δική σας υποστήριξη. Θέλουμε να υποστηρίξουμε και το European Institute of Technology για την επόμενη φάση δραστηριοτήτων. Για το ranking θέλετε να πω κάτι ή με απειλείτε με το σφυράκι σας θα κατανοήσατε την πρόταση αξιολόγησης ranking που προβάλλουμε. Δεν μιλάμε για καταλόγους ή γεράρχηση 1 με 10. Θα πρέπει να συγκρίνουμε ομότιμα, όχι δηλαδή το MIT με κάποιο περιφερειακό πανεπιστήμιο σε μια άκρη της Ευρώπης. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια πρωτίστως και όχι ανταγωνισμός. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν κάνει πράγματα τα οποία βάσει της συνθήκης δεν επιτρέπεται να τα κάνει καθόλου. Αυτό το, το βρίσκω εξαιρετικά καλό. Χαίρομαι που η Κομισιόν προσπαθεί προσπαθεί να εξηγήσει και να προβάλλει το ότι η διακυβερνητική προσέγγιση της Μπολόνια δεν ήταν σωστή και να διορθώσει και πραγματικά καταβάλει τρομερή προσπάθεια να μπορέσει να διορθώσει τα κακό σκήμενα. Και η Μπολόνια δεν θα μπορούσε να είχε πραγματικά ε, να προοδεύσει, να εξελιχθεί, εάν δεν είχαμε χρησιμοποιήσει τα θεσμικά όργανα. Λοιπόν, Ξέρουμε όλοι τα κακό σκήμενα, ξέρουμε τα σφάλματα, έχουμε κυριολεκτικά ε, καταβάλει τεράστιες προσπάσεις να τα ξεπεράσουμε και βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα και από την ε, πολεμική Προεδρία του Συμβουλίου και από την Κομισιόν θα μας ε, διευκολύνουν στο έργο μας να προχωρήσουμε όλοι μαζί για την επόμενη γενιά. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα για την επόμενη γενιά φοιτητών όχι μόνο ε, για τους μαθητές ε, σήμερα, αλλά και για όσους θέλουν να προχωρήσουν στα πανεπιστήμια. Δεν μπορούν όλα αυτά να οργανωθούν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Η, τα πανεπιστήμια ήδη ε, πρέπει κάπου να ρυθμίσουν το θέμα του bachelor, έτσι. ούτε αυτό είναι δύσκολο ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν μια τεράστια κρίση παγκόσμια αλλά και ευρωπαϊκή, άρα πρέπει να είναι πολύ ευέλικτα τα πανεπιστήμια στις προσεγγίσεις τους. Ε, χάρηκα πάρα πολύ για αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα. Πιστεύω ότι γενικά δεν υπήρχαν διαφωνίες. Συμφωνούμε όλοι για το κοινό καλό. Και στο τέλος αυτής της ακρόασης είμαι λίγαν ικανοποιημένη διότι μάσαμε πολλά. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ το Συμβούλιο και την Κομισιόν δια, διαβρύναμε τους ορίζοντές μας και πιστεύω ότι στις εκθέσεις, στις γνωμοδοτήσεις ε, του κ. Μπερλιγκέρ, καταρχάς και άλλος ένας συνάδελφος τον οποίο θα ανατεθεί μια έκθεση, θα περιλαμβάνονται πάρα πολλά ενδιαφέροντα και νέα στοιχεία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία, ολοκληρώνω την ακρόαση και ρωτάω αν υπάρχει τίποτα υπό τα διάφορα στην ημερήσια διάταξη. πρέπει να αποφασίσετε αυτά τα οποία, να ψηφίσετε αυτά που αποφασίστηκαν στην συνεδρίαση συντονιστών. Στα διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Ευχαριστούμε τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε. Καλή όρεξη. Λίγη